Good morning everybody. meeting. Please take your seats. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ώρα να αρχίσουμε τη συνεδρίαση. Παρακαλώ καθίστε. Περιμέναμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να προσέλθουν οι συνάδελφοι, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε με τη σημερινή μας συνεδρίαση ως προσωρινή πρόεδρος κηρύσω την άνταξη της συνεδρίασης Σήμερα θα εκλέξουμε ε, τους προέδρους και τους αντιπροέδρους, τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους σύμφωνα με το 242 του Κανονισμού, πρώτα θα εκλέξουμε τον ή την πρόεδρο και μετά τους ή τις Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία. Βεβαίως όταν κάποιος κάνει μια δουλειά που του αρέσει, ε, αυτό προκαλεί ικανοποίηση αλλά εάν επιπλέον συνεργάζεται με μια ομάδα ανθρώπων όπως ε, αυτούς με τους οποίους συνεργάστηκα εγώ τα τελευταία δυόμιση χρόνια είναι ακόμα πιο ικανοποιητικό. Συγκινήθηκα. Ε, έτσι, έτσι γίνεται. Οι γυναίκες συχνά εκφράζουν περισσότερα συναισθήματά τους θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία, αυτή την καταπληκτική ομάδα που διευκόλυνε το έργο μου. Λοιπόν, βεβαίως ε, ο αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών ε, είναι το πάθος μου και θα συνεχίσω τον αγώνα αυτό με το ίδιο πάθος όπως και όλα τα μέλη της Επιτροπής μας βέβαια. Είμαι βέβαιος ότι η επόμενη ομάδα θα κάνει πολύ καλή δουλειά και θα συνεχιστεί αυτό το πολύ καλό κλίμα συνεργασίας που υπάρχει. Λοιπόν, Να σας πω επίσης ποιοι είναι οι αντικαταστάτες. Ξέρω ότι στη συνεδρίαση αυτή ε, πρέπει να συμμετάσχουν τα μέλη. Εάν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη εδώ, πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία. Για την ώρα ξέρουμε ότι η κυρία Μποσάν ε, η την κυρία Ντανσίδα από τη Σοσιαλιστική Ομάδα και η κυρία Βόρτ ε, η κυρία Χόνιμπολ. Τώρα από το ΕΛΚ η κυρία Σασταρά ε, αντικαθιστά την κυρία Βόζεμπεργκ και έχουμε άλλη μια αντικατάσταση. Η κυρία Μπέρντερ επίσης ε, αντικαθιστά την κυρία Βοσμίνοβα. Και η κυρία Αρένα, ε, ε, συγγνώμη, αντικαθιστάται από τον κύριο Μπόιζα. Από τον κύριο Μόιζα. Λοιπόν, να επαληθεύσουμε ότι υπάρχει εδώ απαρτία ε, επαρκής ε, συμμετοχή για να μπορέσουμε να περάσουμε τώρα στους υποψήφιους για την Προεδρία. Έχουμε λάβει μια πρόταση από την ομάδα των Σελσών από την κυρία Μπλικεβιτσιούτα. Υπάρχουν άλλες προτάσεις. Δεν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση, οπότε εγκρίνεται ομόφωνα. Η κυρία Μπλικεβιτσιούτα ε, είναι πλέον πρόεδρος της Επιτροπής μας, η κυρία Μπλικεβιτσιούτε. Labą dieną Θα μιλήσω λιθουανικά. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, εκ μέρου όλων την απερχόμενη πρόεδρο, την κυρία Πέρεθ. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και ε, σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην θέση της συντονίστριας που είναι εξίσου σημαντική με αυτή της Προέδρου. Θα ήθελα να πω ότι ελπίζω πραγματικά ότι θα μπορέσουμε να εργαστούμε ομαδικά και ότι θα φέρει αποτέλεσμα η προσπάθειά μας σε όλα τα κράτη-μέλη για ε, τα ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πρέπει να εκλέξουμε τέσσερις αντιπροέδρους. Πρώτη αντιπροεδρία απαρτία υπάρχει. Ε, τα πνευματικά μέλη έχουν καταγραφεί ε, από τη γραμματεία για την πρώτη αντιπρόεδρο λοιπόν έχουμε μία υποψήφιο την κυρία Μπάρμπαρα Ματέρα συμφωνεί με την υποψηφιότητά της αλλά δεν είναι εδώ σήμερα δεν μπορεί να συμμετάσχει στη συνάντησή μας. Θα ήθελα να ξέρω εάν υπάρχουν άλλοι ή άλλες υποψήφιες. Όχι. Στην περίπτωση αυτή επιβεβαιώνουμε διαβοής την κυρία Ματέρα ε, στη θέση της πρώτης αντιπροέδρου. Λοιπόν, τώρα θα εκλέξουμε τον δεύτερο δεύτερη αντιπρόεδρο. Ίδια διαδικασία. Η ομάδα Γκούε έχει υποβάλει την υποψηφιότητα του κυρίου Λόπεζ. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Όχι. Θα επιβεβαιώσουμε λοιπόν ε, την υποψηφιότητα του κυρίου Ζωάπου Μέντο Λόπες διαβοής σας παρακαλώ να έρθετε εδώ στο Προεδρείο κύριε Λόπες τρίτος η τρίτη αντιπρόεδρος έχουμε την υποψηφιότητα της κυρίας Χόνιμπολ από την ομάδα των Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Δεν είναι εδώ σήμερα η κυρία Χόνιμπολ Ε, οπότε θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχουν άλλοι ή άλλες υποψήφοι. Όχι. Διαβοή λοιπόν επιβεβαιώνουμε την ε, υποψηφιότητα της κυρίας Χόνιμπολ, τέταρτη αντιπρόεδρος. Έχουμε την υποψηφιότητα της κυρίας Γιάννα Ζιτνάντσκα από την ECR. Δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Ε, Γιάννα, ε, η υποψηφιότητά σου ε, γίνεται αποδεκτή διαβοής και καλείσαι και εσύ να έρθεις εδώ στο Προεδρείο. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής της Προέδρου και των Αντιπροέδρων. Θα πρέπει τώρα βεβαίως να συνεργαστούμε να εργαστούμε ομαδικά και τώρα να περάσουμε στις ε, τακτικές εργασίες μας. Θα πρέπει πρώτα να εγκρίνουμε την εμείς διάταξη. Υπάρχει μια αλλαγή στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για την έκθεση του κυρίου Ορτασούν ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014-2015 ε, αποφασίσαμε το θέμα αυτό ε, τελικά την έθεση γιατί μόνο την ψηφίσουμε στις 6 Φεβρουαρίου και όχι σήμερα. Ωραία, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την σημερινή εμείς διάταξη και τα λοιπά, να την εγκρίνουμε καθώ και τα πρακτικά τη συνεδρίας τη 7 η και 8 η Νοεμβρίου και τη 29 η Νοεμβρίου. Εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά. Τώρα το επόμενο σημείο στην διάταξη θα ψηφίσουμε. Προετοιμαστείτε παρακαλώ. Ε, ε, κοιτάξτε αν έχετε τις κάρτες σας. Λοιπόν, η πρώτη έκθεση επί της οποίας θα ψηφίσουμε είναι η έκθεση της Claire Moody ε, το Ταμείο για την Ισότητα μεταξύ των δύο φύλων ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, σχετικά με το έγγραφο αυτό και τη διαδικασία ψηφοφορία ήθελα δύο σχόλια να κάνω. Ah, e, Έλεγα λοιπόν ότι ήθελα να κάνω δύο σχόλια σχετικά με το έγγραφο αυτό. Τροπολογία 244 και 245. Η πρώτη αναφέρεται στην παρακολούθηση του προγράμματος. το οποίο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2016. Πρόκειται λοιπόν για μια τροπολογία που ε, είναι λαθασμένη υπό την έννοια αυτή. Η 245 αφορά τον προϋπολογισμό του διαμεσολαβητή των δικαιωμάτων του πολίτη στην Πολωνία και εδώ υπάρχει όμως ένα σφάλμα διότι ο διαμεσολαβητής μάλλον ο προϋπολογισμός του διαμεσολαβητή για το 2017 μήπως θα μπορούσα να έχω την προσοχή σας ε, πρόεδρε έλεγα λοιπόν ότι ο προϋπολογισμός του διαμεσολαβητή των δικαιωμάτων του πολίτη στην Πολωνία το 2017 αυξήθηκε κατά 2 εκατομμύρια σλότη. Όμως, στην τροπολογία, οι εισηγητές λένε ότι μειώθηκε ο προϋπολογισμός. Το 2016 ήταν περί τα 35 εκατομμύρια σλότη ο προϋπολογισμός και το 2017 είναι περί τα 37 εκατομμύρια άνω των 37. Επομένως έχουμε μια σαφέστατη αύξηση κατά 2 εκατομμύρια. σλότι. δεν ξέρω από πού βρήκαν τις πληροφορίες οι συνάδελφοι που υπέβαλαν ε, την πρώτη τροπολογία, όμως δεν είναι πραγματικά δεδομένα. Δεν είναι σωστά, εν πάση περιπτώσει. Θα καλούσα λοιπόν την Επιτροπή να καταψηφίσει τις δύο αυτές τροπολογίες, διότι απλούστατα περιέχουν σφάλματα. E, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Βυσνιεύσκα για αυτήν την πληροφορία, το σημειώσαμε. Όμως, καθότι δεν είναι εδώ οι εισηγητές, δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες του περιεχομένου. Όμως, σημειώσαμε την παρατήρησή σας. Και μπορούμε τώρα να περάσουμε στη ψηφορία. Ε, εάν μου επιτρέψετε όμως, ε, Πρόεδρε, 2.44 και 2.45 ήταν τροπολογίες, απλώς να επαναλάβω, τις οποίες ανέφερα. Λοιπόν, ε, η 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 44 είναι σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 48 και 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Τροπολογία 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 72 και 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 75 και 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 82 σε 2, 83 σε δύο τμήματα. Πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 84, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 85, υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 94. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11, συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 117, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 129 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εκατόν τριάντα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ενα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 134. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 135. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 136. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 139 και 141 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται.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 Απορρίπτεται. 153. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 154. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 155. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την 155 ψηφίζουμε. Θα περιμένουμε. Εκατόν λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές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 Ας ελέγξουμε. 164 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Μάλιστα, εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 171 και 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 177 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 178 και 179 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 181 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 183 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 184 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 185 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 186 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 191. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 192. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 193. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 194 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 198 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 199 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ...205 και 206 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 207 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 208 σε μπλοκ μαζί με την 211, 212, 213. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Προϋπολογισμός 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 209. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 214 και 215 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 216 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 217 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 218 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 219 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 220 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 221 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 222 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 224 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Καταπίπτει και περνάμε στην 225. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.26 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Budget 4. Προπολογισμό 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 227. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 228. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 231, 32 και 33. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτονται. 234. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 235. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προπολογισμός 3. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 236 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 237 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 238 Θέλετε να ελέγξουμε την 237. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 238. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προϋπολογισμός 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 242. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κόντ 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 244 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.45. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. 2.45. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Απορρίπτεται. Συγγνώμη. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται. Τροπολογία 6 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20. Υπέρ. Κατά. αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 και 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Budget age. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 και 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Budget D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κόντ G. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κοντ H υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και κοντ I υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε το τελικό ψήφισμα ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Yes, please, Mrs. Vishnevska, the floor is... Κυρία Βυσνιεύσκα, παρακαλώ. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, όλα τα μέλη της Επιτροπής που καταψήφισαν τις τροπολογίες 2.44 και 2.45. Και εκπλήσωμε που υπάρχουν μέλη που θεωρούν ότι μπορούν να ψηφίζουν κατά τρόπο απολύτως παράλογο. Σας είπα προηγουμένως τα μεγέθη, τα 37 εκατομμύρια σλότη του προϋπολογισμού ένταντι των 35 που είναι αύξηση, είναι σαφέστατη αύξηση του προϋπολογισμού, δεν μπορούμε να θεωρούμε λοιπόν ότι το αντίστροφο συνέβη. Σας είπα ξεκάθαρα ότι αυξήθηκε ο προϋπολογισμός διαμεσολαβητή στην Πολωνία, λυπούμε, λυπούμε που ε, οι ιδεολογικές τοποθετήσεις ε, υπερβαίνουν την πραγματικότητα. E, e, Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Πάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο. τη σύσταση στο Συμβούλιο σχετικά με την κατάσταση της γυναίκας. Κωνστάς Μαγκρίτ και... και Μαρία Αρένα. Τροπολογία προφορική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 και 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Όχι. Ναι, ναι, η 51 είχε καταπέσει. Ζητώ συγγνώμη. 36 ε, λοιπόν, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 και 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56, η συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά εποχέ εγκρίνεται 64 υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται 69 υπέρ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 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 και 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται και ψηφίζουμε για το σύνολο άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ πέρασε εγκρίθηκε σας ευχαριστώ Yes, next. Θα προχωρήσουμε τώρα Σχέδιο γνωμοδότησης 2015 απαλλαγή ε, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ε, για την ισότητα των δύο φύλων. κύριε Νταντσίλα είναι συγκεκριμένη. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ, κατά,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 Ναι. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Και εδώ σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε επί του συνόλου της ονομοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε εκ μέρους της κυρίας Δαντσίλα. Και τώρα θα ψηφίσουμε το σχεδίο γνωμοδότηση για την απαλλαγή του 2015 Γενικού Προπολογισμού τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάρει κυρία Νταντσίλα. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Σε δύο σκέλη. Πρώτο σκέλο. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο μέρο. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβιβασμός 2. Υπέρ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 Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα επί του συνόλου υπέρ. Ή μάλλον άρχεται ψηφοφορία, συγγνώμη. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 25 υπέρ και 4 κατά. Ευχαριστώ Βερόνικα. Τέλος. Για την συνεργατική οικονομία. Ανιέσκα Κοσλόφσκα Ράιεβιτς είναι η συγκήτρια. Τροπολογία 3. Υπέρ. Μπορούμε να τα ψηφίσουμε όλα μαζί. Όχι.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Ε, σας ευχαριστώ που ήσασταν τόσο ενεργοί κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Τώρα πρέπει όμως να συνεχίσουμε. Λοιπόν, θα τροποποιήσουμε κάπως την ημέρησια διάταξη τη σημερινή θα ακούσουμε την παρουσίαση του προγράμματος εργασιών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Είναι εδώ μαζί μας η Διευθύντρια αυτού του Ινστιτούτου που θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασιών του έτους 2017 η Βιρτζίνια. Παρακαλώ.

Tai mes tęsiam posėdį ir prašau gerbiamą direktorę Virginiją pristatyti. Συνεχίζουμε λοιπόν τι εργασίε μα. Η Βιτζίνια Λάντμπεργκ έχει το λόγο που θα μας μιλήσει για το πρόγραμμα εργασιών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου και των Σώτο Δύο Φίλων. Το πρόγραμμα του 2017. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ το μέλη του Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, είναι παράδοση ευχάριστη να ξεκινούμε μια συζήτηση εδώ στην Επιτροπή σας για τις πολιτικές προτεραιότητες ε, και τις ανάγκες ε, ε, του Κοινοβουλίου, διότι εσείς μαζί με το Συμβούλιο και την Κομισιόν καθορίζετε και το δικό μας έργο. Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποιες σκέψεις για το προηγούμενο έτος, το 2016. Και τι έφερε για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων το έτος αυτό έχουμε μια αργή πρόοδο. Και υπάρχουν επίσης τεράστιες αποκλήσεις από χώρα σε χώρα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των κανόνων των ευρωπαϊκών και των ε, ε, οδηγιών. Το 2016 είχαμε επίσης κοινωνίες όλο και πιο διαιρεμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε αυτό αφορά το στήμα της μετανάστευσης, της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης ή της ε, υπεράσπισης των παραδοσιακών αξιών. Το θέμα των, της όρης μεταξύ των δύο φύλων συχνά οδήγησε σε πολιτική αντιπαράθεση, ε, σε διέρεση. Οι κοινωνικές ανισότητες και ο αποκλισμός ε, είναι στο επίκεντρο αυτών των κοινωνικών αλλαγών και αυτό δεν είναι τυχαίο ε, και βεβαίω αυτό επηρεάζει και τις βασικές μας αξίες και την ίδια τη δημοκρατία μας. Το θέμα της στόχης παραδείγματος χάρη, αν σας δώσω κάποια παραδείγματα, να σας δώσω κάποια παραδείγματα από τα ευρήματά μας. Βλέπουμε ότι την περασμένη δεκαετία δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως προ... ε, πρόοδος τη μείωση των ισοτήτων σε ό,τι αφορά ε, τις ε, ε, απολαβές. Σε κάποιες χώρες μάλιστα έχει αυξηθεί ε, το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών. Στη Λιθουανία, στη χώρα που βρίσκεται το Ινστιτούτο, είχαμε μια αύξηση των ισοτήτων 7 φορές. Το 2016 εξετάσαμε εμείς ε, ε, την οικονομική κατάσταση στα κράτη-μέλη της Ένωσης ε, υπό το πρίσμα όμως της μεταξύ των δύο φύλων. Να σας δώσω λοιπόν ε, κάποια στοιχεία από την τελευταία μελέτη για την φτώχεια και τις ανισότητες με βάση το φύλο. Εδώ βλέπετε ότι οι οικογένειες με παιδιά έχουν υψηλότερα κίνδυνο φτώχειας. Γιατί, Γιατί οι γυναίκες έχουν λιγότερες πιθανότητες να εργαστούν. Όσο περισσότερο, ε, όσο περισσότερα παιδιά έχουν υπό τη φύλαξή τους, μόλις 55% των γυναικών με τρία περισσότερα παιδιά εργαζόταν το 2015 και από στατιστικής πλευράς όσο περισσότερα παιδιά έχει μια γυναίκα τόσο πιο πιθανό είναι να μην εργάζεται και αυτό βεβαίως έχει σημαντικές επιπτώσεις ε, στη ζωή της. Οι άνεργες γυναίκες είναι πιο ευάλωτες σε αυτά που μπορούν να τους συμβούν. Ε, χωρισμός, ε, θάνατος του σύζυγου, ε, εάν χάσουν το εισόδημα του ε, συντρόφου τους, αυτές και τα παιδιά τους έχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο, διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο να βρεθούν ε, σε μια κατάσταση ένδυας. Ό,τι αφορά τώρα την εκπαίδευση, ε, δεν είναι πλέον η απασχόληση ε, η μόνη συνταγή για να βγει κανείς από την ε, φτώχεια. Η παγκοσμιοποίηση, οι τεχνικές, η τεχνική πρόοδος δημιουργούν νέες μορφές απασχόλησης και νέο περιεχόμενο στις απασχόλησης αυτής. Μετά από αίτημα της Μαλτέζικης Προεδρίας εξετάσαμε ε, την θέση των ε, ανδρών και γυναικών σε ευάλωτες θέσεις εργασίας ε, λόγω χαμηλών δεξιοτήτων ή λόγω χαμηλού εκπαιδευτικού επίπεδου, ε, μορφωτικού επίπεδου. Αν δείτε λοιπόν εδώ την διαφάνεια αυτή θα διαπιστώσετε ότι οι γυναίκες πιο συχνά βρίσκονται, έχουν πιθανότητα μάλλον να βρεθούν σε, μη, σε κατάσταση μη εργασίας. Για να έχουμε λοιπόν μια ορθή λειτουργία της ε, αγοράς εργασίας αλλά και των συστημάτων ε, κοινωνικής πρόνοιας πρέπει να υπάρχει μια εξορρόπηση. Ε, αν δούμε λοιπόν εδώ τι γίνεται με τις δεξιότητες. Ε, αν δούμε τα άτομα με χαμηλές δεξιότητες, ε, βλέπετε ότι η δεξιότητα, η έλλειψη δεξιότητας μάλλον είναι ε, ένας βασικός λόγος για την ανεργία ή για την επισφαλή εργασία μόλις 23% ε, των ε, γυναικών με χαμηλές δεξιότητες ε, από τα 25 έως τα 64 εργαζόντουσαν και μόλις 37% εξ αυτών έχουν επισφαλείς θέσεις εργασίας και μεταξύ των νέων το ποσοστό των, χα... ανδρών με χαμηλές δεξιότητες είναι υψηλότερο από ότι αυτό το γυναικών. Εδώ είναι πολύ ορατό το χάσμα και στις μεγαλύτερες ηλικίε, ιδιαίτερα ναι, στην φάση πρώτης αντισυνταξιοδότησης. Τώρα, για να επιστρέψει κάποιος στην αγορά εργασίας μετά από, ένα, από μια διακοπή, είναι πολύ πιο δύσκολο για τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και χαμηλές δεξιότητες. Αν δείτε εδώ αριστερά τις δύο στήλε ε, με τις χαμηλές δεξιότητες, άντρες και γυναίκες, ε, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες λόγω των διαρθρωτικών ανισοτήτων και των στερεοτύπων τα μισό το 49% αυτών των γυναικών με χαμηλέ δεξιότητε βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας. είναι μόλις 27% το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών. Επιπλέον, εάν δείτε τα στοιχεία αυτά, ε, ε, διαπιστώνουμε ότι έχουμε πάνω από 6 εκατομμύρια γυναίκε με χαμηλέ δεξιότητε και μόλις 2 ε, εκατομμύρια άντρε ε, οι οποίοι δεν, είχαν ποτέ, δεν έχουν ποτέ εργαστεί και πολλοί από αυτού δεν ψάχνουν καν οι περιορισμένες δυνατότητες ε, απασχόλησης ε, ε, επηρεάζουν την απόφαση να εισέλθει κάπου στην αγορά εργασία, ιδιαίτερα όταν η αναζήτηση θέση εργασίας ή ακόμα και η αποδοχή ε, μια θέση εργασία ε, τους αποκλείουν από μια σειρά άλλα επιδόματα και βοηθήματα. Και για τις επισφαλείς θέσεις εργασίας εδώ φαίνεται η διαφορά, ιδιαίτερα σε σχέση με την, ε, με τις απολαβές. Εδώ, αν δείτε τον πράσινο κύκλο, αριστερά, υπάρχει μια σημαντική, μια απόκληση ανάμεσα στα δύο φύλλα. Κάθε πέντε, ένας πέντε άντρες και ένας, μια στις πέντε γυναίκες μάλλον και ένας στους δώδεκα άντρες ε, έχουν πολύ χαμηλές απολαβές και, όταν, και αυτές οι χαμηλές απολαβές έχουν ε, ένα πραγματικό εμπόδιο για την οικονομική ανεξαρτησία και αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερο κίνδυνο να βρεθεί κάποιο στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Αν δείτε τώρα το πιο ε, ροζ κύκλο εδώ για τις, ε, μικτα, τα, τις λίγες ώρες εργασίας, τη μερική αποσχόληση, ε, ε, δεν είναι οι ίδιοι λόγοι για του οποίου οι άντρε και οι γυναίκες ε, δέχονται mini jobs. Ε, πολλοί το κάνουν, πολλές γυναίκες το κάνουν για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Ε, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών είναι πολύ χαμηλότερο. Να σας πω τώρα τι θα κάνουμε φέτος, το 2017. Τα πιο σημαντικά στοιχεία. Βεβαίω το θέμα τη όντω των δύο φύλων δεν είναι ο μόνο τρόπο να φτάσουμε τα ζητήματα αυτά, αλλά ε, είναι και μέρο τη λύση. Ε, χρειάζονται συνολικότερα μέτρα για να υπάρξει μια εξισορρόπηση, να υπάρξει μεγαλύτερη ισότητα. Το να επενδύσουμε δηλαδή στο θέμα τη ισότητα των δύο φύλων ε, συμβάλλει στην ε, απασχόληση, συμβάλλει και στην ανάπτυξη. Και αυτό δείχνει μια πρόσφατη μελέτη, ε, ή μάλλον θα γίνει μια μελέτη φέτος για τα οικονομικά ωφέλη της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Ε, δεν μπορώ να σας δώσω ακόμα τα στοιχεία. Ε, είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα, δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα η μελέτη, έχει γίνει. Η μόνη, η μόνη διαφάνεια που σας δείχνω εδώ δίνει μια εικόνα ε, και δείχνει πως η βελτίωση ευρεία κλίμακας του θέματος των δύο φύλων σε διάφορα επίπεδα μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ έως το 2050 έως και 10%. Πάμε τώρα στο επόμενο, στον επόμενο κλάδο, στο επόμενο πεδίο, σε ό,τι αφορά την πλατφόρμα του Πεκίνου, την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου, ε, έχουμε ασχοληθεί με το θέμα της βελτίωσης των, των δεξιοτήτων των ανδρών και των γυναικών στις επισφαλείς θέσεις εργασίας. Πρόκειται για ένα σημείωμα το οποίο περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα και στοιχεία εν ώψη της Εσθονικής Προεδρίας ε, θα ασχοληθούμε με το θέμα ε, της εκπαίδευσης ε, και των διακρίσεων μεταξύ των δύο φύλων, πώς οι, οι διακρίσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης επηρεάζουν πιο μακροπρόθεσμα και τον χώρο εργασία και την απόκληση απολαβών μεταξύ των δύο τα λοιπά. Τώρα υπάρχει το θέμα της βίας Βεβαίως, η βία παραμένει ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα και συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δράσεις ε, για να πάψει η βία κατά των γυναικών. Θα συμφωνείτε όλοι και όλες μαζί μου ότι ισότητα μέχρι των δύο φύλων η, η απάλληψη των ισοτήτων είναι ένα σημείο κλειδί για να μειωθεί και η βία κατά των γυναικών. Έτσι λοιπόν ε, θα έχουμε το πρώτο πλαίσιο που θα μετράει την βία κατά των γυναικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα μιλήσουμε για τις ρίζες του κακού, ε, για τις αιτίε και το πώς ε, αυτές αναπαράγουν τη βία και τη διατηρούν. Θα προσπαθήσουμε να προσμετρήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Ελπίζουμε ότι αυτό το πλαίσιο μέτρησης, αυτός ο δείκτης ευρωπαϊκός θα, θα βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα να παρακολουθήσει ε, τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, η διάσκεψη του Ισταμπούλ, τα δικαιώματα των θυμάτων, ε, καθώς και ε, η εισαγγελική διαταγή. Ολοκληρώνουμε μια σημαντική και χρήσιμη μελέτη και για το θέμα της ορολογίας να μπορέσουμε να αναρμονίσουμε δηλαδή τους ορισμούς ε, για το θέμα του βιασμού, το θέμα ε, της ε, ε, δολοφονίας γυναικών, δολοφονίας του συζύγου, της συζύγου. Εάν δεν έχουμε τον ίδιο ορισμό για το τι σημαίνει βιασμός, δεν μπορούμε να κάνουμε και συγκρίσεις, διότι καθένας μιλάει για διαφορετικά πράγματα. Αυτοί οι ορισμοί λοιπόν είναι έτοιμοι και θα προσπαθήσουμε να τους προωθήσουμε, συνεργαζόμαστε και με την Στάτη γι' αυτό, για να έχουμε ενιαία, ενιαίους ομόφωνους ορισμούς. Ε, επίσης θα πρέπει να συνεχίσουμε να εκτιμούμε το ποσοστό ε, της κλειτοδιροκτομής, κλειτοδιροκτομής συγγνώμη, ε, είναι κάτι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα με το μεταναστευτικό ζήτημα. Να δούμε λοιπόν πως αυτά τα δικαιώματα των κοριτσιών που κινδυνεύουν θα μπορέσουν να προστατευθούν. Θα εξετάσουμε και την ανάλυση της, δικαι... οδηγίας για την, ε, τα δικαιώματα των θυμάτων από το, υπό το πρίσμα της εμπορίας ανθρώπων. Τώρα περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Όπως βλέπετε, Εδώ εξετάζουμε πώς μπορούμε να μετρήσουμε τη βία κατά των γυναικών ή και τη βία γενικότερα. Βεβαίως τα επίσημα στοιχεία, τα οποία δεν είναι πολλά, αλλά αυτά έχουμε σε επίπεδο Eurostat και από τα εθνικά, σε εθνικές αστικές υπηρεσίες, αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε στο δεύτερο επίπεδο, δηλαδή τα διοικητικά στοιχεία. Ε, πριν από αυτή τη συνάντηση, αλλά και μετά, ε, θα οργανώσουμε συναντήσεις με, με κάθε κράτος μέλος, με τις αστυνομικές αρχές, τις δικαστικές αρχές, για να συζητήσουμε τι μπορεί να συμβεί, πώς μπορούμε να εναρμονίσουμε την συλλογή των δεδομένων, των διοικητικών, για να μπορούμε από εκεί πέρα να τα χρησιμοποιήσουμε για να μετρήσουμε τουλάχιστον τη βία, την ενδοοικογενειακή, ε, καθώς ε, και τους βιασμούς και τους, ε, τις δολοφονίες γυναικών για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα στοιχεία από τις αστυνομικέ και δικαστικέ αρχές θα μπορούμε να τα συλλέξουμε σε όλα τα κράτη-μέλη. Και τώρα να περάσω στο gender mainstreaming. Ένα μακροπρόθεσμο μέρος, ε, μόνιμο μέρος των εργασιών μας. Εμείς ξεκολουθούμε να υποστηρίζουμε την πλατφόρμα για το gender mainstreaming που χρησιμοποιείται σε πέντε μελών ε, από τους ειδικού, τους εμπειρογνώμονες αλλά και από τις κυβερνήσεις και θα επεκτείνουμε αυτή την πλατφόρμα, θα την επικαιροποιούμε σε όλους, σε όλους τους τομείς με νέα στοιχεία ε, το θέμα της όντως των δύο φύλων και της εκπαίδευσης. Υπάρχει μια μεγάλη μελέτη για να δούμε πώς ε, ε στον τομέα της εκπαίδευσης ε, μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο μας στα πλαίσια της Μαλτέζικης Προεδρίας, θα αναλύσουμε τις πτυχές που έχουν να κάνουν την ισότητα των δύο φύλων στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συμβαίνει και τώρα για να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους, να βρούμε τους κατάλληλους δείκτες, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το σύστημα. Θα ήθελα επίσης με την ευκαιρία να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το σχετικό δίκτυο για το Gender Mainstreaming για το ενδιαφέρον και τη συνεργασία που είχαμε έτσι να προχωρήσουν οι εργασίε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Εμείς ε, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Τώρα για το gender budgeting. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητούμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε πολλές περιπτώσεις ε, έχουμε καταλάβει ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην, στην Επιτροπή σας. Ε, τώρα πρέπει να αποφασίσουμε βεβαίως για ποιο, ποιο διαθροτικό ταμείο θα μπορούσε να αναλύσει ε, σε βάθος το ζήτημα για να προετοιμάσουμε κάποιες τελευταίες γραμμές, κάποια προσέγγιση, να δούμε από τα διαφορετικά ταμεία της Ένωσης ποιο θα μπορούσε να είναι πιο χρήσιμο για αυτή την απόπειρα ε, να υπάρχουν κάποιες δημοσιονομικές γραμμές για την θεματισότητα των δύο φύλων, για το gender budgeting. Τέλος. Βεβαίως, ε, όπως πάντα και φέτος, ε, γύρω στον Οκτώβριο θα έχουμε την τρίτη έκδοση του δίκτυ για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, του index. Όχι μόνο θα επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία, θα δούμε τι συμβαίνει από το 2005 έως σήμερα, ε, πώς πάει αυτή η τάση μείωση των ισοτήτων, ε, υπάρχει μείωση. Ε, επίσης θα έχουμε το πλήρες πλαίσιο που θα αφορά την βία κατά των γυναικών με βάση τα δεδομένα που θα έχουμε στη διάθεσή μας και βεβαίως θα πρέπει να δούμε τις, ε, τις ανισότητες ε, τις οριζόντιες ε, θα πρέπει να μπορούμε να προσμετρήσουμε κάποιες από τις παραμέτρους τις σχετικές πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον έχουμε προσθέσει και κάποιες νέες μεταβλητές στον τομέα της υγείας στην οποία επικεντρωνόμαστε όλο και περισσότερο, καθώς και στον τομέα της ε, εξουσίας ε, σε κοινωνικό επίπεδο. Θα τα δείτε όλα αυτά τον Οκτώβριο ε, και ελπίζω να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτό έτσι εντάχει για τα στοιχεία με τα οποία ασχολείται, τα στοιχεία που συλλέγει το Ινστιτούτο έτσι ώστε από εκεί πέρα οι, οι πολιτικές αποφάσεις να παίρνονται περιστατωμένα. Προσπαθούμε να παίξουμε ένα ρόλο για να δίνουμε στοιχεία που έχουν να κάνουν με το σε όλα τα επίπεδα ε, πολιτικής της Ένωσης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και βεβαίως ε, αναμένω να συνεχιστεί η συνεργασία μας. Ευχαριστούμε. Την κυρία Λάνμπακ, ε, λέει πρόεδρος. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το λόγο, αλλά ευχαριστώ ακόμα περισσότερο για την παρουσίασή σας. Γνωρίζουμε όλοι το έργο που κάνετε, το έργο που κάνει το Ινστιτούσιο για την Ισότητα των Φύλων, που δίνει αποτελέσματα, προσπαθεί να συλλέξει στατιστικά στοιχεία, τα οποία νομίζω επιβεβαιώνουν ε, το προέστημα που έχουμε. Πολλοί εδώ στην Επιτροπή Γυναικών έχουμε μία εικόνα, μία αίσθηση του τι κάνετε, όμως αυτά είναι πραγματικά τα στοιχεία που το αποδεικνύουν. Γι' αυτό με εκπλήσει κάθε φορά που μας φέρνετε νέα στοιχεία, ε, τα οποία πάλι επιβεβαιώνουν τους φόβους μας πολλές φορές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για την ε, τακτική ενημέρωση. Μία ερώτηση έχω να κάνω. Μας ε, είπατε πώς συλλέγετε δεδομένα αριθμούς εδώ και πολλά χρόνια, αλλά συγκεκριμένα η βία ε, κατά των γυναικών, η ακροδεξιά βία, πώς επηρεάζει τις ε, γυναίκες, υπάρχει κάποια αλλαγή, υπάρχουν κάποια, κάποιες παράμετροι οι οποίες πρέπει να υπολογιστούν εκ νέου έτσι ώστε να μετρήσουμε ε, σωστά τα ποσοστά της βίας. Υπάρχουν επίσης ορισμένες πόλεις οι οποίες παρουσιάζουν αυξημένη τέτοια βία κατά των γυναικών. Ε, υπάρχει δηλητηριασμένη ατμόσφαιρα για τις γυναίκες, για τα δικαιώματα των γυναικών. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω αν εσείς έχετε κάποια συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία για να... που θα ρίξουν φως στο τι συμβαίνει ακριβώς σε αυτά τα μέρη. Τι έχετε διαπιστώσει, ποιες είναι οι παρατηρήσεις που κάνετε και τι γίνεται με την άφηξη των νέων ε, στην Ευρώπη, προσφύγων, μεταναστών, πώς αλλάζουν εκείνοι την ε, κατάσταση, τη ζωή των γυναικών σε αυτές τις ε, πόλεις και των γυναικών που έρχονται και των γυναικών που βρίσκονται ήδη εδώ και τι μπορούμε να αναμένουμε τα επόμενα 5 ή 10 χρόνια. Ε, μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη βασισμένη στα δεδομένα που έχουμε. Νομίζω πως και για μένα προσωπικά αλλά και για πολλούς συναδέλφους τα στοιχεία που συλλέγετε και επεξεργάζεστε είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί με αυτά Μπορούμε να ε, περιγράψουμε τα φαινόμενα που χαρακτηρίζουν την κοινωνία που αλλάζει. Thank you Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε είναι ε, να συλλέγουμε δεδομένα. Τα δεδομένα που αφορούν τη βία κατά των γυναικών σπανίζουν. Και αυτό που λέτε κι εσείς, ε, το να εξετάζουμε πόσο συχνά απαντώνται αυτά τα φαινόμενα, ε, ναι, με, μας δίνει κάποια εικόνα, όμως δεν είναι και η ακριβής πραγματικότητα. Τώρα, υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο εξετάζουμε τα δεδομένα, τα εξετάζουμε ποσοτικά, ε, αλλά προσπαθούμε πάντα να έχουμε και ένα ποιοτικό πλαίσιο. Προσπαθούμε να έχουμε και το συγκείμενο και το υπόβαθρο όλων αυτών των δεδομένων που συλλέγουμε. Γι' αυτό λοιπόν και αυτή τη στιγμή ε, έχουμε τα αποτελέσματα της ε, μελέτης που κάναμε και σχεδιάζουμε τη συνέχεια. Έχουμε εστιάσει στους μετανάστες, ιδιαίτερα στο εκπαιδευτικό σύστημα και ορισμένες προκλήσεις που εσείς αναφέρατε, που αφορούν τις αξίες, τον ε, εκφοβισμό των γυναικών, τη βία. Θεωρούμε πως τα δεδομένα που συλλέγουμε θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να διεξάγουμε κάποιες αναλύσεις για το τι γίνεται με τους μετανάστες, πώς ε, γίνεται η ένταξη των ε, μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα, πώς μπορούμε να υπερασπιστούμε ε, τις γυναίκες και πώς ε, αλλάζει η νέα σύσταση του, των σχολείων το εκπαιδευτικό σύστημα. όπως γνωρίζετε ενδεχομένως, η στα αυτή τη στιγμή εξετάζει αυτόν τον επιπολασμό, έτσι ώστε να μπορούμε εμάς, να, εμείς μετά να επιβεβαιώσουμε, αν θέλετε, αυτές τις ε, τάσεις που διαφαίνονται από τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα. Μετά, ε, αυτά τα διοικητικού τύπου δεδομένα αφορούν ε, δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από τις αρχές επιβολής του νόμου, από το, το σύστημα δικαιοσύνης, από την αστυνομία. Αυτά αποτελούν μέρος του όγκου των δεδομένων και Φυσικά είναι δεδομένα που χρειάζονται επεξεργασία. Φέτος σκοπεύουμε να συνεχίσουμε με αυτή την ανάλυση έτσι ώστε να καταφέρουμε να διακρίνουμε τις διαφορές στα κάθε κράτος μέλος και να δούμε πώς η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η πρόληψη θα λειτουργήσει με το βέλτιστο δυνατό τρόπο σε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά η ισότητα των φύλων είναι στον πυρήνα όλων των προσπαθειών. Γι' αυτό λοιπόν και χρειάζεται να γίνει πολύ καλή και εντατική δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο θα πάρει η κυρία Γκαρσία Περές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Λάνμπακ για την παρουσίασή της ε, και την τακτική της επαφή με την ε, Κομισιόν. Θεωρώ ότι πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής μας και του Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων, διότι και για εμάς ε, πρόκειται για ένα μέσο που ενισχύει τη δουλειά σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορα βήματα. Στο πρόγραμμα που έχετε σχεδιάσει για το 2017 υπογραμμίσατε διάφορα θέματα επί των οποίων θα εστιαστούν οι μελέτες σας ε, και που σχετίζονται και με πολλές από τις γνωμοδοτήσεις που εμείς έχουμε προγραμματίσει. Θεωρώ λοιπόν ότι θα είναι πολύ σημαντική αυτή η επαφή. Όπως είπε και η κυρία Νόχιλ, υπάρχει μια ανησυχία που εκφράζεται την Επιτροπή, δηλαδή να είμαστε σε θέση να ποσοτικοποιήσουμε σε όλες αυτές τις στατιστικές μελέτες με ποιον τρόπο υλοποιούνται τα βήματα αυτά. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και ενώσεις ε, ε, γυναικών σύλλογοι, μη όμικρον, ε, έχουν, αναπτύσσουν την εντύπωση ότι υπάρχουν βήματα προς τα πίσω. Ε, στην όλη προσπάθεια της ισότητας του φίλου, στην ε, αναπαραγωγική σεξουαλική πρακτική, στην ε, εκπαίδευση των παιδιών, το σύνολο της δουλειάς που μπορεί να βάλει στο τραπέζι το Ινστιτούτο σχετικά με την πραγματικότητα που αισθάνεται και που εκφράζει η κοινωνία των πολιτών θα είναι πολύτιμο για εμάς για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε ε, τις εκκλήσεις μας προς τα θεσμικά όργανα της Ένωσης ε, και προς τα πολιτικά κόμματα. Ευχαριστώ. Yes, also... Ναι. Διαβάζοντας τα διάφορα σχέδια γνωμοδοτήσεων ε, και εμάς μας ικανοποιεί ιδιαίτερα ότι χρησιμοποιείται όλο και περισσότερα στοιχεία από τη δουλειά μας τα οποία προσπαθούμε να επικαιροποιούμε το συντομότερο δυνατό, το συχνότερο δυνατό. Τακτικά κάνουμε και μια παρακολούθηση, έχουμε και μια νέα τράπεζα δεδομένων και πολύ συχνά μπορούμε να αντλήσουμε τα δεδομένα ακόμα και χωρίς εκθέσεις. Πράγματι και εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι η ποστικοποίηση, η δυνατότητα της ποστικοποίησης είναι πολύ σημαντική. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κυρία Ρένκεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι συνάδελφοι ήδη εξέφρασαν τις ευχαριστίες προς εσάς και σας ευχαριστώ και εγώ. Μιλήσατε για τις διαφορές μεταξύ των κοινωνιών, την, το σχετισμό με τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, και εμείς έχουμε δει τα προβλήματα αυτά, αλλά ήθελα να πάω σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Νομίζω ότι η απειλή ε, προς τα δικαιώματα των γυναικών είναι και λόγω μιας, ε, αν θέλετε, πολιτιστικής αντίδρασης που εκφράζεται αυτή τη στιγμή ε, και λόγω του ευάλωτου χαρακτήρα των ανδρών και της αρσενικότητας έτσι όπως εκφράζεται από τις κοινωνίες μας ο δυνατός τύπος που κερδίζει το ψωμί για τον οικοκυριό και που ενδεχομένως κάθε τόσο ε, χειροδική κιόλας. Πρέπει να δούμε τις πολιτιστικές τάσεις και αλλαγές που έχουμε στην κοινωνία και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε ή να επηρεάσουμε αυτά τα πρότυπα της αρσενικότητας του ανδρισμού. Εμείς ε, προφανώς και πιέζουμε για να επικυρωθεί η σύμβαση της Ισταμπούλ και ήθελα να ξέρω αν έχετε δεδομένα αναλυτικά από τα κράτη-μέλη σχετικά με το ποια κράτη έχουν επικυρώσει και ποια δεν έχουν επικυρώσει τη σύμβαση. Και σε σχέση με τον ορισμό του βιασμού αλλά εσεί θεωρείτε ότι η επικύρωση τη σύμβασης θα είχε σημαντικό αντίκτυπο από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τελικώ και από πλευρά όλων των κρατών μελών. Κοιτάξτε, λέει η κυρία Λάνμπακ, ε, σχετικά με το ευάλωτο του χαρακτήρα του ανδρισμού και αυτά που αναφέρατε, ναι, είναι πράγματι υφίστανται όλα αυτά. Εμείς συμπεριλαμβάνουμε τις πτυχές αυτές σε όλες μας τις μελέτες και όπως αναφέρθηκα και στην μελέτη σχετικά με την ε, παιδεία και εκεί θα είναι σαφέστατο. Διότι η μελέτη αυτή βασίζεται στην ε, διακήρυξη του Παρισιού σχετικά με τις τάσεις αυτές και θα έλεγα προς το τέλος του φθινοπόρου θα έχουμε περισσότερα συγκεκριμένα στοιχεία και με χαρά θα τα μοιραστούμε μαζί σας. Θα έχουμε επίσης και την παρακολούθηση των ζητημάτων των σχετικών με τη μετανάστευση που θα είναι και αυτό ένα κομμάτι που θα πρέπει να προσθεθεί. Αλλά αυτό το φαινόμενο του ευάλωτου ανδρισμού διατρέχει διάφορους ε, τομείς αν θέλετε. Είναι οριζόντιας φύσεως. Έχουμε και αυτήν την εκστρατεία White Ribbon, που και αυτή είναι μια προσπάθεια καταπολέμησης της βίας, και είναι μια προσπάθεια επιρροής των ανδρών ώστε να γίνει μια συζήτηση και νομίζω ότι και σε επίπεδο κρατών μελών ε, υπάρχουν δράσεις και πριν από το συνέδριο της Μάλτας έχουμε την υψηλού επίπεδου συνάντηση σχετικά με τους άντρες, αν καταλάβαμε καλά την ομιλήτρια. Ε, σχετικά με την επικύρωση τώρα της σύμβαση. έχουμε κάποια δεδομένα περισσότερο για δική μας χρήση. Γιατί περισσότερο δουλεύουμε με οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, για παράδειγμα. Για εσωτερική μας χρήση, λοιπόν, έχουμε κάποια τέτοια δεδομένα. Δεν κάναμε follow-up γιατί έχουμε πολλή δουλειά με τις βιστάμενες τρέχουσες μελέτες. Αλλά όταν θα έχει ολοκληρωθεί η προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης στη, στην σύμβαση, θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η παρακολούθηση από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τότε θα έχουμε τα πλήρη δεδομένα, τους ορισμούς όπως είπατε, όπως και τα διοικητικά μεγέθη. Θα είναι λοιπόν αν θέλετε, επίσημα σε εκείνο το σημείο και σε εκείνο το σημείο θα μπορέσουμε να συνεισφέρομαι. Σας ευχαριστώ κυρία Μίλνερ. Ε, άλλη μία ερώτηση και από πλευρά μου. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω τα όσα είπε συνάδελφος. Αυτού του είδους η παρακολούθηση θα βοηθήσει, θα ενισχύσει τα επιχειρήματά μας, ελπίζοντας και πιστεύοντας ότι θα έχουμε και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα το θέμα της σύμβασης στρέφεται και προς την ε, Προεδρία και όλοι ανησυχούμε σχετικά με το ρόλο της Πολωνίας στο πλαίσιο αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε περισσότερες πληροφορίες. Και όπως ελέγχθη και εγώ θα επιβεβαίωνα ότι έχει κανείς την αίσθηση μιας αντίδρασης ιδιαίτερα ακούγοντας ε, δηλώσεις ε, εκλεγμένων προέδρων ή ηγετών από διάφορες χώρες. Επίσης, δεν ξέρω αν έχετε πληροφορίες σχετικά με την ε, άρση των, της απαγορεύσεως των αμβλώσεων γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν τρία σημεία όπου εστιάζεται το lobbying ε, προς τα μέλη του Κοινοβουλίου ότι σχετίζεται με τα δικαιώματα των ζώων, την Παλαιστίνη και το Ισραήλ και τα σεξουαλικά δικαιώματα, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Σε οτιδήποτε άλλο είμαστε πολύ μακριά από τα επίπεδα πιέσεως σε αυτά. Επομένως αν έχετε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θα μας ήταν πολύτιμη. Κοιτάξτε, για τη σύμβαση και για περιπτώσεις τύπου Πολωνία. Αυτό είναι περισσότερο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς χρειαζόμαστε πλήρης αποδείξεις, πλήρη στοιχεία. Βεβαίως και έχουμε επαφές και συζητήσεις αλλά δεν βρίσκεται στον έλεγχό μας το πράγμα. Ε, σχετικά τώρα με τις απαγορεύσεις ε, των αμβλώσεων και τα σχετικά αναπαραγωγικά δικαιώματα και εκεί πράγματι βλέπουμε ένα αντίστροφο κύμα, ένα κύμα αντιδραστικό και πρέπει να αναλύσουμε τα στοιχεία για να δούμε ποια είναι τα πιο ισχυρά μας επιχειρήματα. Εκεί υπάρχουν και οι συγκρούσεις των δικαιωμάτων, τα δικαιώματα της γυναίκας, τα δικαιώματα του παιδιού. Πρόκειται για περίπλοκα ζητήματα βέβαια, επί των οποίων εμείς δεν εργαζόμασταν γιατί ήταν και θέματα των κρατών μελών. Δηλαδή υπάρχουν και διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και εμείς ε, μπορούμε να δουλεύουμε μόνο επί θεμάτων επί των οποίων υπάρχει συνένεση για τα κράτη-μέλη. Και σε αυτό το ζήτημα δεν έχουμε συνένεση όπως γνωρίζετε, αλλά είναι πράγματι πολύ σημαντικό να έχουμε ε, ενιαίες προσπάθειες, κοινέ προσπάθειες από όλους τους φορείς και θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η, η κυρία Ward. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και για την παρουσία και την εκπρόσωπο του Ινστιτούτου και για τη δουλειά που έχετε κάνει, η οποία είναι πολύτιμη για μας. Και σας ευχαριστούμε που υποβάλλετε ποσοτικά δεδομένα, αλλά βέβαια όλοι ξέρουμε ότι πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται άνθρωποι. Και η δική μας δουλειά είναι να συσχετίσουμε ακριβώς τους ανθρώπους αυτούς, τους αριθμούς αυτούς με τους αριθμούς. Και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, είτε είναι οι γυναίκες που υφίστανται βία, είτε είναι ε, ομάδες πληθυσμού που πλήττονται από τη λιτότητα. Ε, η δική μας δουλειά είναι να υποβάλλουμε και να υπογραμμίζουμε αυτά τα ζητήματα. Διερωτώ με κατά πόσον καταφέρατε να συλλέξετε δεδομένα σχετικά με φαινόμενα πολιτικής βίας, κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με ανησυχεί όλο και περισσότερο. Η Τζο Κόξ στο Ηνωμένο Βασίλειο δολοφονήθηκε όπως θα ξέρετε λόγω των του πολιτικών της πιστεύω. Επομένως δεν μιλούμε μόνο για πολιτική βία σωματική αλλά και πολιτική βία που ασκείται μέσω διαδικτύου στη δημόσια σφαίρα, στα μέσα επικοινωνίας και είναι κάτι το οποίο ε, πλήττει ακόμα περισσότερο τις γυναίκες και μάλιστα τη στιγμή που χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες εκπροσώπους παρά λιγότερες. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερα δεδομένα σχετικά και με τέτοια φαινόμενα για να μπορέσουμε να τα φέρουμε στο προσκήνιο με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Πράγματι, λέει η κυρία Λάνμπακ, είναι ένα φαινόμενο με αυξητική τάση. Εμείς δεν έχουμε εστιάσει συγκεκριμένα επί της ε, πολιτικής βίας. Αλλά στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και στο πλαίσιο του Πεκίνου υπό την ε, Λουξιμβουριανή Προεδρία είχαμε μία σχετική ανάλυση η οποία δεν ήταν πλήρης γιατί έπρεπε να εστιαστούμε και περισσότερο σε άλλες περιοχές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μερικώς καλύπτουμε το θέμα αυτό στο νέο εργαλείο που έχουμε αναπτύξει από πέρυσι στην Διακοινοβουλευτική Ένωση και για το πόσο ευαίσθητα είναι τα διάφορα εθνικά κοινοβούλια απέναντι στα ζητήματα της ιστότητας των φύλων Έχουμε, έχουμε αναπτύξει κάποιους δείκτες για το πόσο ενθαρρύνουν τα κοινοβούλια με τη δράση τους τα θέματα αυτά. Και νομίζω ότι ένας από αυτούς δείκτες συνδέεται και με το περιβάλλον, λέει ο Μιλήτρια. Και εν των επομένων εκλογών, λέει ομιλήτρια, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ακόμη πιο σημαντικό το θέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναγκάζομαι να πάρω το λόγο, διότι οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στην Πολωνία, τη χώρα μου. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα σχόλια είναι βία κατά κάποιο τρόπο. Στην Πολωνία έχουμε μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, στηρητική, η οποία είναι κατά των εκτρώσεων και υπέρ της ζωής. Πρέπει να το σεβαστείτε αυτό. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί διαμαρτύρεστε. Εγώ είμαι συντηρητική. Βαθιά συντηρητική. Και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να εξωστρακιστούμε. Έχουμε κάθε δημοκρατικό δικαίωμα να είμαστε υπέρ τη ζωή. Υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία Πολωνών που θεωρεί ότι η ζωή είναι ιερή και πρέπει να προστατεύεται από τη στιγμή τη σύλληψη. Ήμουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 2004-2005 είχα μιλήσει για το θέμα αυτό Και εγώ θέλω να αλλάξω ε, την, ε, τον ορισμό της ε, αναπαραγωγικής υγείας. Δεν είμαστε ζώα που απλά κάνουμε αναπαραγωγή. Εγώ θέλω να μιλήσω ε, για procreation και όχι για reproduction. Μόνο τα ζώα αναπαράγονται. Θα ήθελα λοιπόν να, να σας ζητήσω να σεβαστείτε τη δημοκρατική μας απόφαση. Δεν είμαστε τίποτα άγριοι που δεν έχουμε ακόμα εκπολιτιστεί κάναμε την επιλογή μας. Υπάρχουν πολλές απόψεις. Κάποιοι θεωρούν ότι κάποιος που έχει κάνει έκτρωση ε, είναι τραυματισμένος μετά, ως το θάνατό του. Ε, θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τις γυναίκες που είναι έγκυες και δεν θέλω να νιώθω ότι στιγματίζομαι και ότι εξωστρακίζουν εδώ. Παρακαλώ, η συνάδελφος. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Νόχλη, που μου δίνετε το λόγο αμέσως, γιατί δεν μπορώ να αφήσω την απάντησή μου να περιμένει. Ε, ναι, έχετε κάθε δικαίωμα να πρεσβεύετε τη γνώμη σας ε, και φυσικά έχετε κάθε δικαίωμα να πιστεύετε πως η κυβέρνηση της Πολωνίας εκπροσωπεί την πλειοψηφία του πολωνικού λαού. Η δικαίωμά μου είναι όμως να έχω και τη δική μου άποψη, να την εκφράζω ελεύθερα, να έχω και, την άποψη, και το δικαίωμα να εκφράζω την άποψή μου ελεύθερα για το τι κάνουν οι άλλες χώρες και πώς ε, αυτό επηρεάζει. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ε, έχω να πω ότι ε, με προσβάλλει αυτό που λέτε. Εμείς ε, δεν προσβάλλουμε κανέναν, δεν επιτιθέμεθα σε κανέναν και εγώ προσωπικά πιστεύω πως είναι απαράδεκτο για την κυβέρνηση της Πολωνίας να νομίζει πως μπορεί να αποφασίσει για τις ζωές και τα δικαιώματα όλων των γυναικών. Και το πλήθος των γυναικών που κατέβηκε στους δρόμους να διαδηλώσει την Πολωνία το αποδεικνύει. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Ward. Ναι, αν δεν, έχω, αν δεν κάνω λάθος, η μεγάλη κινητοποίηση στους δρόμους της Πολωνίας γυναικών και ανδρών λόγω της πρότασης περιορισμού της έκτρωσης στην Πολωνία απέτρεψε την κυβέρνηση από το να πάρει αυτό το μέτρο. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι υπάρχει κάποια δράση από τα κάτω, υπάρχει κάποια αντίδραση από τα κάτω και αυτό έρχεται τώρα να γενικευθεί με τις ε, ε, πορείες των γυναικών ανά τον κόσμο λόγω της εκλογής του Πρόεδρου Τραμπ. Ε, όλο και περισσότερες γυναίκες από διαφορετικό, διαφορετικά περιβάλλοντα ενθαρρύνουν να συμμετάσχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες. Μιλήσατε για βία με έναν περίεργο τρόπο. Λες και αυτό που κάνουμε εδώ, εδώ στις εργασίες μας στο Κοινοβούλιο ε, έχει κάτι να κάνει με τη βία. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι αυτοί που ε, αναζητούν εκτρώσεις μη νόμιμες, τότε αυτοί είναι τα πραγματικά θύματα μιας βίας, μιας τραγικής βίας από μη ασφαλείς εκτρώσεις και έχουμε πάρα, πολλές, πάρα πολλούς θανάτους ε, και παιδιών ε, και γυναικών επειδή οι γυναίκες σε αναψώμενες χώρες δεν έχουν την κατάλληλη περίθαλψη. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα Ινστιτούτο το οποίο να συλλέγει στοιχεία για να έχουμε εμείς εμπεριστατωμένα δεδομένα για να μπορέσουμε να καθορίσουμε τις πολιτικές μας. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι που το επιθυμούσαν πήραν το λόγο, έθεσαν τα ερωτήματά τους θα ήθελα εγώ ε, να ζητήσω η συνεργασία της Επιτροπής μας με το Ινστιτούτο ε, να συνεχιστεί αλλά έχω και ένα ερώτημα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς έτσι ώστε αυτή η συνεργασία έτσι ώστε όλες αυτές οι μελέτες να είναι προσβάσιμες σε όλες τις υπόλοιπες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι είναι δύσκολο να αποδείξει κάποιος ότι η ισότητα των δύο φύλων είναι σημαντική όταν παίρνονται αποφάσεις σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε αυτό, το πώς δηλαδή αυτές τις πληροφορίες θα διαδοθούν τα αποτελέσματα των μελετών σας παραδείγματος χάρη Και κάτι άλλο. Όταν εξετάζουμε τι γίνεται στους 28 κράτη-μέλη, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλές αποκλίσεις από χώρα σε χώρα. Και πολλές αποφάσεις εξαρτώνται από τις πολιτικές προσωπικότητες, αντιπροσωπικότητα των πολιτικών ηθινόντων στις χώρες αυτές και πρέπει εμείς να είμαστε ενωμένοι. Πρέπει να εξηγούμε γιατί η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων είναι χρήσιμη σε όλους τους τομείς. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τη Βιργίνια Λάνμπακ, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, που βρίσκεται στη Λιθουανία. Είμαι, είμαι και εγώ Λιθουανή και ελπίζω να συνεχιστεί η συνεργασία μας με τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο νομίζω πως ε, ο καλύτερος τρόπος ε, για να διαδώσουμε τις πληροφορίες στις άλλες επιτροπές ε, είναι να περάσουμε από εσά, διότι μιλούμε με διάφορους κλάδους άλλους μας λένε τι σχέση έχει αυτό με το δύο φίλων έχουμε πολλά εργαλεία, έχουμε πολλά δεδομένα και επιχειρήματα ε, και αυτός νομίζω πως είναι, το καλύτερο για φέτος οι άλλες επιτροπές δηλαδή να ε, μάθουν να ε, αντιληφθούν πως η πολιτική ισότητα των δύο φίλων επηρεάζει το δικό τους τομέα πολιτικής. Ευχαριστώ για τη συνεργασία. Ministrė, tuoj ateis, todėl mes turbūt turim kokių penkių penkių. Κυρία e, Υπουργέ, από τη Μάλτα, η, υπουργό Υπουργός μάλλον της Μάλτας έχει αργήσει, θα έρθει σε λίγα λεπτά, οπότε ένα μικρό διάλειμμα πριν έρθει η Υπουργός Κοινωνικού Διαλόγου της Μάλτας. Gerbiami kolegos, mes mūsų posėdį. Αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Συνεχίζεται λοιπόν η συνεδρίαση και σήμερα έχουμε προσκεκλημένη στην Επιτροπή την Υπουργό της Μάλτας για Κοινωνική Προστασία προστασία των καταναλωτών κοινωνικού διαλόγου. Κυρία Μαρινεταλή, θα μας παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Μαλτέζικης Προεδρίας στον τομέα των δικαιωμάτων της γυναίκας, της ισότητας των φύλων. Κύριε Υπουργέ, σας δίνω τώρα μέσω στο λόγο. Okay. Καλημέρα σας κύριε, και κύριοι. Για τα τελευταία 60 χρόνια η Ευρώπη θεωρούταν ένας φάρος ειρήνης, ανάπτυξης και ευημερίας. Αυτά όλα όμως αποκτήθηκαν σε μια εποχή όπου πολλοί αμφεβαλάνε ότι θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε. Στην 60η επέτειο του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος είναι η σειρά της Μάλτας, του μικρότερου κράτους μέλους, να ε, αναλάβει αυτήν την τιμή της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια εποχή όπου μαζί πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό των τελευταίων 60 ετών. Όλοι έχουμε υποχρέωση να ε, προστατεύσουμε όλους και να ε, πληροφορήσουμε τους πολίτες, να τους μεταδώσουμε ε, τα ωφέλη που έχουν αποκτήσει τα τελευταία 60 χρόνια και που πολλές φορές κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία που με τα χαρά θα αναλάβουμε να εκπληρώσουμε. Η Ευρώπη χρειάζεται νέα ορμή και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ήπειρό μας δείχνουν ότι υπάρχει μια σαφής ανάγκη για την Ευρώπη να έρθει πιο κοντά στους πολίτες της και να επικοινωνεί μαζί τους με αποτελεσματικό τρόπο, να τους ενημερώνει για, ε, τις, ε, για το, αυτά που προσπαθεί να κάνει για εκείνους, για όφελος των πολιτών και για τα όσα κάνει προσπαθώντας να κάνει τους πολίτες να επιτύχουν τους στόχους τους. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει εμπειρίες που θυμάδεψαν όλους μας και η ανάγκη για μεταρρύθμιση ποτέ δεν ήταν πιο επιτακτική. Γι' αυτό λοιπόν περισσότερο από ποτέ πρέπει να έρθει ο ένας πιο κοντά στον άλλο. Τα γεγονότα του τελευταίου έτους συγκλώνησαν το, τα θεμέλια του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και η Μάλτα είναι αποφασισμένη να συνεισφέρει θετικά στην Ευρώπη. Ελπίζουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας με τη δουλειά που θα κάνουμε στο Συμβούλιο και με εσάς, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταφέρει να εξέλθει πολύ δυνατότερη από αυτήν την κρίση. Γνωρίζουμε βέβαια ότι είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα των έξι μηνών, αλλά έχουμε την ε, φιλοδοξία να καταφέρουμε πολλά μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα και να διασφαλίσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πιο αξιόπιστη. Γνωρίζουμε τους περιορισμούς και τις ελλείψεις μας, αλλά γνωρίζουμε και τα δυνατά μας σημεία. και στο Συμβούλιο θα παρουσιαστούμε με ειλικρίνεια, χωρίς ε, κρυμμένη ατζέντα, χωρίς ε, προσπίτη ευγένεια. Γι' αυτό λοιπόν αυτό θα το μεταφέρουμε και στο Κοινοβούλιο και ελπίζουμε αυτό το πνεύμα ειλικρίνειας και συνεργασίας να αποδώσει καρπούς ο Πρωθυπουργό ε, και όλο το επιτελείο της κυβέρνησης αλλά και οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης έχουν διατελέσει μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό νομίζω είναι μια απόδειξη του πόσο γνωρίζουμε τη δουλειά που γίνεται εδώ και πόσο την ε, αξιολογούμε. Είμαστε λοιπόν υπερήφανοι για το ότι ήρθε η σειρά να αναλάβουμε αυτή τη χρονική στιγμή την Προεδρία του Συμβουλίου. Οι κύριες αρχές που διέπουν την Προεδρία μας θα ε, είναι να δώσουμε μία νέα όθηση στην Ευρώπη, να φέρουμε τους πολίτες πιο κοντά ως καταναλωτές, ως ε, πολίτες που παράγουν πλούτο και ως... Ε, σημαντικού ε, φορεί. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε εντοπίσει έξι τομεί προτεραιότητα: Τη μετανάστευση, την ασφάλεια, την ενιαία αγορά, την ευρωπαϊκή γειτονία, ε, κοινωνική συμπερίληψη και ε, ζητήματα ναυτιλίας. Είναι πολύ σημαντικό, διότι οι πολίτες μας έχουν σοβαρές ανησυχίες τις οποίες πρέπει να εισακούσουμε και νομίζω πως κάθε προτεραιότητα πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά. Γι' αυτό, με την άδειά σας, κυρία Πρόεδρε, θα αναφερθώ στη δουλειά που θα κάνουμε στο πρόγραμμα της ε, Μαλτέζικης Προεδρίας σε αυτούς ε, τους τομείς που αφορούν τη δική σας Επιτροπή. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Γυναικών, τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή σας και το Κοινοβούλιο ήταν πραγματικά φάρος ελπίδας για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα. Αυτή η εποχή ζητά ισότητα και έχουμε δει όλοι όσοι ασχολούμαστε με την ισότητα σε καθημερινή βάση ότι ο πυρήνας στη κοινωνική ψυχή της Ευρώπης αποτελείται ακριβώς από την ισότητα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθεί ένας διάλογος με τον καθημερινό άνθρωπο, την καθημερινή γυναίκα και να καταφέρουμε με αυτόν τον τρόπο να συνδέσουμε τους πολίτες με αυτά που κάνει η Ευρώπη, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι μας. Έχουμε πολεμήσει για την ισότητα των φύλων κατά της βίας ε, εναντίον των γυναικών και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Εγώ προσωπικά με την ιδιότητά μου ως υπουργό ε, συνεχίζω τις προσπάθειες και θέλω να εκφράσω την ευχαρίστησή μου που υπάρχει η ευρωπαϊκή δέσμευση να εξαλειφθεί οποιαδήποτε μορφή έμφυλης βίας. Το καλύτερο εργαλείο που έχουμε είναι η Σύμφαση της Κωνσταντινούπολης και χρειάζεται λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι όσο το δυνατόν περισσότερα ε, κράτη θα επικυρώσουν τη σύμβαση αυτή. Η Προεδρία της Μάλτας έχει υποσχεθεί να θέσει το ζήτημα αυτό στους ε, υψηλότερους στόχους και στις υψηλότερες προτεραιότητες. Γι' αυτό λοιπόν και θα γίνει μια συνέντευξη τύπου για την έμφυλη βία που πλήττει κυρίως στις γυναίκες, όπου θα γίνει και μια έκκληση για καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ας μην ξεχνάμε ότι στην επικράτεια της Ένωσης μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί κάποια μορφή βίας τουλάχιστον μία φορά στη ζωή της. Επομένως, η απαλυφή αυτής της μορφής βίας απαιτεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία συμπεριλαμβάνει πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες από πλευράς κρατών μελών, καταρχάς για να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα, η ποιότητα και η αξιοπιστία των δεδομένων, να ε, συνεχίσει η ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσω εκστρατιών, να υπάρχει καλύτερη στήριξη στα θύματα της έμφυλης βίας, να ε, φροντίσουν έτσι ώστε η δικαιοσύνη να ε, κάνει το έργο της ε, για όσους κριθούν ένοχοι και ε, να σταθώ τώρα στο εξή. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τον σεξισμό αλλά και τον ρατσισμό, την ομοφοβία, την τρανσφοβία και άλλες διασυνδόμενες μορφές διακρίσεων η εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων ήταν για πολλά χρόνια ένα βασικό ζήτημα που απασχολούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Προεδρία της Μάλτας αναγνωρίζει το πόσο σημαντική είναι η συγκεκριμένη πρόταση και υπόσχεται λοιπόν να προσπαθήσει να προχωρήσουν οι συζητήσεις σε αυτό το κεφάλαιο. Μόνο μέσω ενός συντονισμένου καθιερωμένου ευρωπαϊκού κοινοτικού πλαισίου θα διασφαλίσουμε πως οι γυναίκες θα εκπροσωπούνται επαρκώς στα θεκητικά συμβούλια των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών. Η Προεδρία μας επίσης αποσκοπεί στην ε, στην ε, εφαρμογή της νέας πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την ε, εξισορρόπηση της κατάστασης στα δύο φύλλα, έτσι ώστε να πρέπει προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα για να μπορούν και οι εργαζόμενες γυναίκες να ε, έχουν μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την οικογενειακή και προσωπική ζωή. Αυτή η πρωτοβουλία που έχουμε κατά νου θα έχει θετικό αντίκτυπο στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, δεδομένων των ε, στοιχείων που έχουμε που ε, απαιτούν αυτή τη συμφιλίωση εργασίας, μητρότητας και προσωπικής ζωής. Η Προεδρία της Μάλτας δεσμεύεται για την ε, επιθυμητή ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή. Όλες οι γυναίκες έχουν δικαίωμα και να κάνουν οικογένεια, αλλά ταυτόχρονα ε, και να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Πρέπει λοιπόν να επιτευχθεί η ισορροπία ανάμεσα στα δύο. Γι' αυτό η Προεδρία μας θα ε, προσπαθήσει όσο καλύτερα μπορεί να ε, ακολουθήσει αυτόν τον ε, στόχο βασισμένη στην ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Προεδρία μας επίσης έχει κάποια συμπερά... βασίζεται σε κάποια συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις γυναίκες που εργάζονται σε επισφαλείς θέσεις ή που έχουν χαμηλά ή ελλειπή προσόντα. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλέ γυναίκες αλλά και άντρε που συναντούν μεγάλες δυσκολίες στην επανένταξή του στην αγορά εργασίας. Τώρα, ε, σε ό,τι αφορά τις ίσες ευκαιρίες για συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας, ε, να πω πως εξακολουθεί να είναι ένα προβληματικό ζήτημα. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο πολιτικής, για παράδειγμα το Σύμφωνο για την ε, Ισότητα, την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για μια στρατηγική ε, που θα στοχεύει στην ισότητα. Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε δείχνουν ότι η αγορά εργασίας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις στον τομέα αυτών αντιμετωπίζουμε αυξανόμενο κίνδυνο ε, επισφαλών θέσεων απασχόλησης ε, τις οποίες καταλαμβάνουν γυναίκες και οι γυναίκες με χαμηλά προσόντα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να παραμείνουν άνοιγες από ότι οι άντρες. Η επανένταξη τώρα ε, ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας είναι ένας από τους ε, στόχους μας. Η Προεδρία της Μάλτας θα συνεχίσει να εργάζεται στον τομέα της ισότητας και θα επεκταθεί το, η προσπάθεια αυτή σε πολλούς τομείς. Ε, πέρα από την προσπάθεια για απαλληφή της έμφυλης βίας και το σχετικό συνέδριο στις 2 Φεβρουαρίου, η Προεδρία μας θα ε, φιλοξενήσει και το, και το Υπουργικό Συμβούλιο για τους ε, ΛΟΑΔ. Προβλέπεται το συνέδριο αυτό να λάβει χώρα στις 23 Φεβρουαρίου και θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να δοθεί δημοσιότητα στην ισότητα των φύλων και να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο ε, πάνω στα συμπεράσματα του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν το 2016 τον Ιούνιο αλλά και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, ισότητα σε θέματα ΛΟΑΔ. Επίσης, η Προεδρία μας θα γιορτάσει την Παγκόσμια ημέρα κατά της ομοφοβίας με διάφορες εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες της Βρυξέλλης. Η Προεδρία μας επίσης θα αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες που αφορούν το φύλλο σε διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερα, για παράδειγμα, το Μάρτιο στο Διεθνές Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Γυναίκες. Όπως σας είπα και πριν, η Μαλτέζικη Προεδρία έχει ως προτεραιότητα ε, την συζήτηση για την έμφυλη βία. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να το τονίσουμε ε, καθ' όλη τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, Ευχαριστούμε την Υπουργό για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Μαλτέζικης Προεδρίας για τα θέματα της ισότητας των φύλων. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τους ε, συντονιστές να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, τις ερωτήσεις τους. με Κοράσα, παρακαλώ εκ μέρους της Κωνσταντ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε Υπουργέ για τα σχόλια σας. Ε, στο ΕΛΚ ε, είμαστε δεσμευμένοι για την προώθηση των θεμάτων ισότητας των φύλων, καταπολέμησης των διακρίσεων και της ενίσχυσης θέσης των γυναικών ε, στη ζωή και στην επαγγελματική σταδιοδρομία με ίσες ευκαιρίες χαιρόμαστε που εστιάζεστε στα θέματα βίας γιατί και εμείς θέλουμε να εστιαστούμε στα, σε εκείνα τα ζητήματα που μπορούμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη συνένεση και στήριξη. Χαιρετίζουμε και τα σχολεία σας για τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης καθότι είμαι και η εισηγήτρια σχετικά με την ε, επικύρωση, την προσχώρηση της Σύμβαση Επομένως ε, πρέπει να ε, καταφέρουμε να επηρεάσουμε τα πράγματα και για τα κράτη-μέλη που δεν έχουν προσχωρήσει και για να προχωρήσει το θέμα της επικύρωσης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει, υπάρχουν αντιρρήσεις σχετικά με τον ορισμό του φύλου και εδώ είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε τι λέει το Συμβούλιο της Ευρώπης και τι λέει η Σύμβαση. η σύμβαση λέγει ομιλεί για βία που ασκείται κατά της γυναίκας μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκα. Πρέπει λοιπόν να διευκρινίσουμε, να αποσαφηνίσουμε αυτή τη διαφορά. Δεν έχει καμία σχέση με χριστιανικές αξίες, αρχές ή οικογενειακές αξίες το θέμα. Επίσης ε, έχουμε δεσμευτεί στο ΕΛΚ ε, και απέναντι σε άλλες μορφές βίας κατά των γυναικών σεξουαλικής ε, παρενόχλησης και κακοποίησης από τους ε, εμπόρους, ε, τους λαθρεμπόρους ανθρώπων. Έχουμε επισκεφθεί κέντρα προσφύγων στην Ελλάδα, στην Τουρκία και αλλού με άλλα μέλη συναδέλφους και έχουμε εγκρίνει και ένα ψήφισμα για ασφάλεια για τις γυναίκες καλύτερους, ε, καλύτερες υγειονομικές συνθήκες ε, και η εστίασή σας επί των ε, γυναικών μεταναστών και προσφύγων υπό την έννοια αυτή είναι πολύτιμη. Η παρακολούθηση των συστάσεων αυτών και του ψηφίσματος είναι επίσης πολύ σημαντική για μας. Θεωρούμε ότι και η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, όπως και εσείς είπατε, είναι ένα ζήτημα κλειδί για τα θέματα ισότητας. Πρέπει να ενισχύσουμε την γυναική επιχειρηματικότητα με συγκεκριμένες δράσεις. Ίσως μισθός για ίδια εργασία είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα για εμάς. Όπως και σωστή πρόσβαση στις ε, υπηρεσίες υγείας εγώ ως πρώτη αντιπρόεδρος της ΣΥΜΚΟ θα πρέπει να πάω εκεί τώρα και ζητώ συγγνώμη που θα απουσιάσω. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Γκαρθία Πέρι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ την Υπουργό εξ ονόματος ε, της ομάδας των Δημοκρατών και Σοσιαλιστών να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, για την παρουσίασή σας επίσης, ε, στην οποία είδαμε πολλά από τα ζητήματα να υπογραμμίζεται που και εμείς επεξεργαζόμαστε καθημερινά. Φακέλους που αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτοί ή στην Κομισιόν, στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο και ήθελα να σας διαβιβάσω την αγανάκτηση της Επιτροπής απέναντι στην έλλειψη πολιτικής στήριξης σε ζητήματα, σε φακέλες που θα περιμέναμε να έχουμε στήριξη από το Συμβούλιο ιδιαίτερα, ιδιαίτερα όπως στην οδηγία στην οποία αναφερθήκατε. Αυτή η συνένεση που θα έπρεπε να υπάρχει και που ελπίζουμε η Μαλτέζικη Προεδρία να μπορέσει να προωθήσει ήθελα να σας ζητήσω να καταβάλλετε όλες τις προσπάθειες ώστε να έχουμε μια κοινή θέση που να μας επιτρέψει να διαπραγματευτούμε. Κατανοούμε ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις, αλλά η ανάγκη του να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, να συζητήσουμε προκειμένου να φτάσουμε σε συμφωνίες είναι θεμελιώδης. Δεν μπορεί να διατρέχονται η μία προεδρία την άλλη και να υπάρχει απόλυτη ε, έλλειψη ικανότητος να λάβουμε, να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία. Επομένως, πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να συνεργαστούμε ώστε να προωθήσουμε το φάκελο αυτό, όπως και στα θέματα της συμφιλίωσης, εμείς είχαμε εγκρίνει μια προκαταρκτική γνωμοδότηση για να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει με τις προτάσεις των τομέα αυτών που πρέπει βεβαίως να εξετάσουν διάφορα θέματα αλλά είναι ουσιαστική σημασία να έχουμε νομοθετική πρόταση εδώ σε αυτό το πεδίο γιατί αυτό είναι τελικά εκείνο το οποίο επιτρέπει και στα κράτη-μέλη να προχωρήσουν. Και όταν αποσύρθηκε η πρόταση οδηγίας ε, για την άδεια μητρότητος, ε, άφησε ένα νομοθετικό κενό. Επομένως, εάν η Προεδρία σας προωθήσει ενεργά αυτά τα θέματα, οπωσδήποτε εμάς θα μας ε, βρείτε στο πλευρό σας, ώστε να ασκήσουμε την επιρροή και την πίεση που μπορούμε στην Κομισιόν για να προχωρήσουν τα θέματα αυτά. Όπως επίσης ε, είπε και η κυρία Κοράσα, ε, δουλέψαμε στα θέματα της ε, βίας, ε, στα θέματα των ε, μεταναστών και των προσφύγων. Είχαμε υποβάλει και γνωμοδότηση από την Επιτροπή μας και την περασμένη εβδομάδα έγινε και συζήτηση στο Κοινοβούλιο που ζητούσε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση απέναντι στα φαινόμενα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στα κέντρα με το κύμα του ψύχους Όλα αυτά είναι σημεία επί των οποίων θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και θα ολοκλήρωνα επαναλαμβάνοντας τη στήριξη που οπωσδήποτε θα έχετε από την ε, Επιτροπή μας αλλά θα σας παρακαλούσα να κάνετε ό,τι είναι δυνατόν ώστε αυτό το μπλοκάρισμα ε, των θεμάτων, η έλλειψη στήριξης πολιτικής των θεμάτων ισότητα των φύλων να τα, μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε. Η επιτυχία θα είναι επιτυχία αυτής της προσπάθειας για εσάς αλλά και για όλη την προσπάθεια της ε, υποστήριξης των γυναικών και της θέσης τους στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε ε, την κυρία Γαρθία Πέρες και κυρία Μίλναρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την Υπουργό που ήταν εδώ μαζί μας και που μας παρουσίασε τις προτεραιότητες ε, του προγράμματος της Μαλτέζικης Προεδρίας. Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που σας περιμένουν στους ερχόμενους έξι μήνες ε, το οποίο το παρουσίασε και στην Ολομέλεια Στρασβούργο ο πρόεδρος σας ήθελα να συμφωνήσω απολύτως ε, με τα όσα είπε η ε, συνάδελφος η κυρία Γκαρθία Πέρες πράγματι έχουμε αγανακτήσει το λέω και προσωπικά αλλά και ως συντονίστρια των θεμάτων της γυναίκας εντός της ομάδας των φιλελευθέρων είναι σαν να ερχόμαστε ξανά και ξανά στο ίδιο θέμα. Ζητούμε κάθε νέα προεδρία ε, να διευκρινίσει, να ξεκαθαρίσει τη θέση της για τη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης και να προχωρήσει το θέμα αυτό. Θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε, δεν πρόκειται να σταματήσουμε, αλλά θα θέλαμε επιτέλους να υπάρξει μια κάποια επιτυχία κάποια στιγμή. Ε, εσείς μπορείτε να υπολογίσετε σε εμά και εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να υπολογίσουμε σε εσά για την προσπάθεια αυτή. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένα τα οποία δεν αναφέρατε και έχω να σας ρωτήσω καταρχάς ποια είναι η στρατηγική της ε, Προεδρίας της Μάλτας ε, για το θέμα του Women on Board και καθότι 1η και 2η Φεβρουαρίου θα έχουμε την ε, συνάντηση υψηλού επίπεδου για το gender mainstreaming. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψή σας ε, να ακούσουμε τι περιμένετε από αυτή τη συνάντηση, από αυτό το συνέδριο εσείς. Ευχαριστώ κυρία Μπιόρκ, τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε και σας καλωσορίζω κύριε Υπουργέ θερμά στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να θέσω κάποια ζητήματα. Κάποια τα ανέφεραν και οι συνάδελφοι. Πρέπει να προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά το θέμα της βίας κατά των γυναικών, το θέμα της επικύρωσης της Σύμβασης της Ισταμπούλ από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τα επιμέρους κράτη-μέλη. Ε, κάτι άλλο τώρα. Η συνεδρία της Κομισιόν ε, για την κατάσταση των γυναικών ε, βλέπουμε ότι ο κύριος Τραμπ δεν χάνει χρόνο ήδη υπέγραψε ένα διάταγμα που απαγορεύει τη χρηματοδότηση ε, όποιων ε, δράσεων υπάρχουν που έχουν σχέση με την έκδοση ακόμα και τις ενημερωτικές θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει δράση άμεσα όπως έγινε και επί ε, διακυβέρνησης Μπούς εμείς ε, πρέπει να καλύψουμε αυτό το κενό, το χρηματοδοτικό το οποίο θα ζήσουν και θα επηρεάσει, και θα επηρεάσει τις οργανώσεις που προσπαθούν να βοηθήσουν τις γυναίκες στις περιπτώσεις αυτές. Ελπίζω λοιπόν να επιδείξετε ε, έτσι ε, ένα ε, πνεύμα επιθετικό στο θέμα αυτό και το Μάρτιο να το δείξετε. Μιλήσατε για το θέμα της ισορροπίας μεταξύ των δύο φίλων Αναμένουμε την πρόσθεση της Κομισιόν βέβαια για του διάφορου ε, διακανονισμού σχετικά με τη γονική άδεια. Εγώ θέλω να θίξω όμω ένα θέμα ε, που ξέρω ότι η Μάλτα ε, τα πάει πολύ καλά. το θέμα τη περίθαλψη των παιδιών, τη φροντίδα των παιδιών, συγγνώμη. Ε, πώς θα μπορέσουμε τους στόχους μας να τους μετατρέψουμε σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο και να το εφαρμόσουμε. Εσείς ε, με την Προεδρία σας θα μπορέσετε να κάνετε τη διαφορά στο θέμα αυτό σε σχέση με τους στόχους ε, για τη φροντίδα των παιδιών. Το τρίτο θέμα που αποτελεί προτεραιότητα για την Προεδρία σας είναι το κοινό σύστημα ασύλου. Στην Επιτροπή μας εξετάζουμε το θέμα ε, των γυναικών προσφύγων η κατάσταση είναι πραγματικά απαράδεκτη. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν νομοθετικές προτάσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε ε, και το θέμα αυτό, το θέμα επίσης των ΛΟΑΤ, το θέμα των παιδιών, όλα αυτά όλες αυτές οι ομάδες είναι ακόμα πιο ευάλωτε στον κόσμο, των προσφύγων. Και κάτι ακόμα. Η Κομισιόν θα υποβάλει μια στρατηγική κατά της, ε, για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Εμείς επικεντρωνόμαστε βεβαίως ε, στο θέμα των γυναικών και των μικρών κοριτσιών εδώ. Πώς μπορούμε εδώ να οδηγηθούμε σε μια στρατηγική που θα επιστιάζει σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Ε, ευχαριστώ Παρακαλώ, επόμενη ομιλήτρια, κυρία Ρένκε, σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και την Υπουργό ε, που μας παρουσίασε το πρόγραμμά της. Ε, οι συνάδελφοι εξέφρασαν ε, την απογοήτευσή τους από τα τελευταία χρόνια απέναντι στο Συμβούλιο, αλλά και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορισμένες φορές. Ένας μισογίνης είναι αυτή τη στιγμή ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ε, εγώ είμαι κάπως πιο αισιόδοξη βέβαια, διότι αν δούμε αυτές τις εξελίξεις αυτό δείχνει ότι πρέπει να παλέψουμε ακόμα περισσότερο για να ακουστεί η φωνή των γυναικών για μια πιο ανοιχτή κοινωνία και ελπίζουμε, ελπίζουμε ότι εσείς θα μπορέσετε να το πράξετε αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν θέλω βέβαια να σας πιέσω, έχετε έξι μήνες, εμείς περιμένουμε αποτελέσματα. Ε, πολλά έχουν ήδη αναφερθεί από τους συναδέλφους, θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία σημεία πιο συγκεκριμένα. Ε, το θέμα των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια πρέπει εδώ να πετύχουμε κάτι. Εγώ κάνω έκκληση εδώ. Ιδιαίτερα η γερμανική κυβέρνηση στη στιγμή το μπλοκάρει το θέμα αυτό. Ε, βασιζόμενοι ουσιαστικά σε ιδεολογικά επιχειρήματα. Οπότε πιέστε τους Γερμανούς συναδέλφους σας παρακαλώ διότι αυτό μπορεί να είναι το σημείο καμπής για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε κάπου στο θέμα αυτό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Το δεύτερο τώρα, επειδή, επειδή αναφερθήκατε στη συνθήκη τη Ρώμη, η οποία ε, ε, υπογράφηκε πριν από 60 χρόνια, λέγονται πολλά και σημαντικά στη συνθήκη αυτή, αλλά υπάρχει μία φράση εξαιρετικά σημαντική. Ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι μια υπόσχεση που δώσαμε πριν από 60 χρόνια και η οποία δεν έχει γίνει ακόμα πραγματικότητα. Επειδή για να αναφερθήκατε επίση στην επισφαλή εργασία, ε, η Επιτροπή μα ε, θέλει πραγματικά να πιέσει έτσι ώστε να υπάρξουν, υπάρξει νομοθεσία για αυτό το σημαντικό θέμα, το θέμα ε, τη ανισότητα σε ό,τι αφορά την αμοιβή, τι απολαυέ. Και κάτι ακόμα που έχει να κάνει με την κυβέρνησή σα και το έργο που έχετε επιτελέσει τα τελευταία χρόνια, έχετε πολύ προοδευτική νομοθεσία για τα διεμφυλικά ζητήματα ε, και επίσης για τα ζητήματα ΛΟΑΤ ε, και τη διάσκεψη που θα οργανώσετε θα μιλήσετε για τα διαφιλικά ζητήματα ε, και τη της Προεδρίας σας θα προσπαθήσετε να προωθήσετε νομοθεσίες ε, πιο προοδευτικές σχετικά με την αναγνώριση των διαφόρων αυτών κατηγοριών και των ιδιωτήτων τους. Ο κύριος Τροτσίνσκι έχει το λόγο, παρακαλώ, η κυρία Τροτσίνσκι. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, ε, τους επόμενους έξι μήνες θα είστε το σημείο αναφοράς ε, για μας, ε, την Επιτροπή Γυναικών. Ε, σημείωσα τις προτεραιότητες που θέλετε εσείς να, να προωθήσετε. Έχω δύο ερωτήματα. Το πρώτο αφορά την πολιτική που ακολουθείται στη Μάλτα από το 2013 και μετά, σε ό,τι αφορά την ισότητα μεταξύ των δύο φίλων και τα ειδικά δικαιώματα για τα άτομα ΛΟΑΤ. Ε, εγκρίνατε μία νομοθεσία gender ε, identity και gender characteristics act που θεωρείται η πιο προοδευτική στην ιστορία. Δικαίως, ε, όντως δίνεται τη δυνατότητα να μπορεί κάποιος να αλλάξει φύλλο κάνοντας μια δήλωση απλά στο Δήμο. Αυτό έχει να κάνει με κάποιο αίτημα ε, της κοινωνίας ε, της Μάλτας ε, ή ήταν ιδεολογική άποψη κάποιας ελίτ ή κάποιον λόμπι και υπάρχουν στοιχεία για το πόσα άτομα χρησιμοποίησαν αυτό το νόμο για να αλλάξουν φύλλο. Επίσης ε, ένα άλλο θέμα που έχει συζητηθεί ιδιαίτερα και πολλοί θέλουν να αποφύγουν, μιλούν απλά για μια διαφορά, γλωσσική. Θέλω να μιλήσω για, το, για την ε, ταυτότητα των φύλων και την ισότητα των φίλων. Σε πολλές εκθέσεις της Επιτροπής δεν μιλάμε για φυσικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μιλάμε για μια ταυτότητα φύλων, όπου πλέον δεν, καθορι, δεν διαχωρίζει άνδρες και γυναίκες ε, από τη φυσική πραγματικότητα, αλλά από την ιδέα που έχει κάποιο τον εαυτό του με βάση τις σεξουαλικές του πρακτικές. Είναι λογικό σε ένα νομοθετικό κείμενο ε, ευρωπαϊκό, το οποίο θέλει να υπερασπιστεί την ισότητα των ανδρών και των γυναικών, να βασιζόμαστε στις σεξουαλικές πρακτικές των ατόμων. Σα ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Υπουργό να απαντήσει στις ερωτήσεις και μετά θα περάσουμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Παρακαλώ. I will answer the questions. Um, Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω στις ερωτήσεις ε, για τις οποίες είμαι αρμόδια και για τις υπόλοιπες θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο μπορώ. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την πρώτη ερώτηση, δηλαδή την καταπολέμηση όλων των μορφών ε, βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Είναι ένα βασικό κομμάτι που αφορά τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και η Προεδρία μας δεσμεύεται να προσπαθήσει για αυτήν την απαλήφη όλων των μορφών της έμφυλης βίας και θα ενθαρρύνει όλα τα κράτη-μέλη να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης όλα τα κρατημέλη, να σας πω, έχουν υπογράψει τη σύμβαση, αλλά όχι επικυρώσει. Η προσχώρηση λοιπόν στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι κάτι που συζητάμε στην αντίστοιχη ομάδα εργασίας του Συμβουλίου και η Προεδρία μας ε, είναι αισιόδοξη για το ότι θα υπάρξει πρόοδος κατά τη διάρκεια της ε, θητείας μας εδώ. Είναι μία από τις ε, κορυφαίες προτεραιότητές μας, γι' αυτό λοιπόν να είστε βέβαιοι πως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ε, τώρα σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, μετανάστες και, την, και το τράφικινγκ. Και αυτό αυτή είναι μια προτεραιότητα της Προεδρίας μας. Τώρα, για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Υπάρχει μια συνένεση για το ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις επιχειρήσεων, αλλά όπως γνωρίζετε υπάρχουν διάφοροι ε, τρόποι να γίνει αυτό. Υπάρχει μεγάλη πολυμορφία, διαφορές στα κράτη-μέλη, υπάρχουν... Υπάρχει διαφορετική πρόοδος από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, αλλά σίγουρα επιδέχεται βελτίωση η κατάσταση. Ωστόσο, όταν το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ συζήτησε το θέμα αυτό το Σεπτέμβριο του 2015, μία ε, μεγάλη μειοψηφία κατάφερε να μπλοκάρει την ε, συνέχεια. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει πρόταση για μία ρήτρα ευελιξίας που θα αφορά κράτη-μέλη τα οποία ήδη έχουν εφαρμόσει μέτρα για να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Θα προχωρήσουμε λοιπόν όσο μπορούμε την ε, συζήτηση στο θέμα αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει συμφιλίωση αυτών των δύο. Γι' αυτό η Προεδρία μας θα χρησιμοποιήσει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα αυτών. Σίγουρα η ισορροπία αυτή είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες όλων των πολιτών, γυναικών, ανδρών, ε, γονέων, παιδιών, εξαρτώμενων μελών της οικογένειας. Είναι πολύ βασικό εδώ να υπάρχει ευελιξία και να σεβαστούμε τις διαφορετικές ε, προσεγγίσεις που προκύπτουν από τις διαφορετικές ε, οπτικές γωνίες των κρατών μελών, αλλά και τις ιδιαιτερότητες από χώρα σε χώρα. Και να λάβουμε υπόψη και την πλευρά των εργοδοτών. Σίγουρα ένα σημαντικό στοιχείο θα ήταν η δωρεάν ε, παιδική μέρημνα και θα προσπαθήσουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τα θετικά παραδείγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που μπορώ να πω μέχρι τώρα είναι ότι τα αποτελέσματα των προσπαθειών είναι πολύ ενθαρρυντικά. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τις προσπάθειες. Τώρα, υπάρχει η σχετική, τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και αυτό που θα κάνουμε είναι να παροτρύνουμε τα κράτη-μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες τους για την σημερινή εκτίμηση της διάστασης του φύλου στην ε, κοινωνική και εργατική πολιτική, να καταρτιστούν σχέδια δράσης που θα καταπολεμήσουν την πρόορη εγκατάλειψη του σχολείου και θα αντιμετωπίσουν τη, αποτελεσματικά τις προκλήσεις που ε, αντιμετωπίζουν αγόρια και κορίτσια που εγκαταλείπουν το σχολείο πρόωρα. Επίσης, ε, θα θέλαμε να δούμε μία αναγνώριση επίσημη αναγνώριση δεξιοτήτων ατόμων που προέρχονται από τρίτες χώρες και έχουν ανάγκη αυτές οι τυπικές ή άτυπες δεξιότητες να αναγνωριστούν. Επίσης, θα προσπαθήσουμε να ασκήσουμε πίεση για την καταπολέμηση της επισφαλούς απασχόλησης και την ε, βελτίωση των συνθήκων εργασίας, παροτρύνοντας τις επιχειρήσεις να λάβουν σχετικά μέτρα που θα οδηγήσουν στην επίτευξη ισορροπίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ε, ΛΟΑΤΚΙ, να σας πω πως ε, θα γίνει ένα συνέδριο στα πλαίσια της Προεδρίας μας, όπου θα γίνει μια παρουσίαση του τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα και όσοι παρευρεθούν στο συνέδριο αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματά τους στο σωστό φόρουμ. Είναι θέμα βέβαια εθνικής αρμοδιότητας ε, όλο αυτό το ζήτημα, αλλά νομίζω πως εκεί θα είναι το, το καλύτερο βήμα για να συζητηθούν τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεύτερος γύρος ερωτήσεων τώρα. Η κυρία Γκάμπριελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας, ε, κυρία Υπουργέ. Καλώς ήλθατε στην Επιτροπή Γυναικών. Ε, θα έχετε οπωσδήποτε τη στήριξή μας, ώστε οι επιθυμίες μας να γίνουν πραγματικότητα για όλες τις γυναίκες στην Ευρώπη, αλλά και πέραν της Ευρώπης. Καταρχάς, ως εισηγήτρια της οδηγίας Women on Board, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που εξέφρασαν τη στήριξή τους, και τη δική μου προσωπικά ως εισηγήτρια για να κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να ξεμπλοκάρουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Το μήνυμα που θέλουμε να διαβάσουμε σε όλες εκείνες γυναίκες που θέλουν πραγματικά να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητε τους πρέπει να είναι θετικό. Ε, επίσης στήριξη από πλευράς μας ώστε να έχετε ένα, το μέγιστο δυνατό αριθμό πρωτοβουλειών ώστε να ασκηθεί επιρροή στα κράτη-μέλη για να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Και μην διστάσετε να χρησιμοποιήσετε και τις, ε, τους μηχανισμούς συντονισμού που έχουμε στη θέση μας γιατί ε, είναι η ανησυχία για αρκετά κράτη-μέλη της εφαρμογής που τα αποτρέπει από την επικύρωση. Και εκμεταλλευόμενοι και την ε, ε, εστίαση της Μαλτέκης ε, Προεδρίας για την Μεσογειακή Λεκάνη, όλα αυτά που κάνουμε για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο είναι υπέρ της ασφάλειας και της σταθερότητας όλων. Και η θέση της γυναίκας ή στην μεσογειακή αυτή λεκάνη, στις ε, βόρειο-αφρικανικές χώρες, ε, στις χώρες του Μαγκρέμπ, έχετε αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να υποστηρίξουμε τη θέση της γυναίκας ε, στην οικονομία και στην παιδεία ιδιαίτερα στον χώρο αυτό. Έχετε προβλέψει κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ευχαριστώ κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί Υπουργέ, όπως βλέπετε υπάρχει πάθος, ενθουσιασμός για τα θέματα αυτά. Γιατί είναι από τα λίγα θέματα από των οποία υπάρχει νομοθετική πρόταση στο τραπέζι και μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Ξέρουμε πως έχουν τα, τα πράγματα στις διάφορες αν θέλετε εθνικές πραγματικότητες Ας μην επιμείνουμε σε αυτό. Ήθελα απλώ να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί σας ε, παρακολούθησα προσεκτικά. Όταν λέτε ότι η Μαλτέζικη Προεδρία είναι έτοιμη να κάνει τα πάντα προκειμένου να βοηθήσει. Να μιλήσει με τη γερμανική κυβέρνηση, με τη σουηδική κυβέρνηση. Γνωρίζουμε, εν πάση περιπτώσει, που υπάρχουν ε, ανησυχίες σε σχέση με προηγούμενε εκλογές, αλλά έχετε προγραμματίσει κάποιο συνέδριο, κάποια εκστρατεία, κάτι το ορατό. Γιατί βλέπετε ότι όλες οι πολιτικές ομάδες είναι έτοιμες να σας υποστηρίξουν, αλλά πολύ συχνά χρειαζόμαστε κάτι που να φαίνεται, που να είναι ορατό. Σας ρωτώ λοιπόν, ως προς τις προτεραιότητες της Προεδρίας τι συγκεκριμένο μπορούμε να κάνουμε. Για το εγγυητικό μέσο των παιδιών, την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια επιμείναμε σε αυτό. Το οποίο βεβαίως όπως γνωρίζουμε συνδέεται με τις πολιτικές ε, ε, ισότιμης μεταχείρισης. Και εδώ έχετε προγραμματίσει κάτι να σας ρωτήσω. Ευχαριστώ. Η κυρία Ward. Ευχαριστώ. Ήθελα να πω κάτι πολύ προσωπικό, οπότε θα περιμένω. Ναι, ε, κυρία Ντάλη, καλώς ήρθατε και εγώ να πω. Σας ευχαριστούμε για την πολύ σταθερή θέση και τοποθέτηση που έχετε για τα δικαιώματα των LGBT LGBTI μάλιστα, και στις διάφορες εκδηλώσεις ε, και στο Pride ε, το πρόσφατο έμαθα ότι είστε ε, ένας πραγματικός φάρος για θέματα ισότητος στην Ευρώπη. Για τα θέματα των δικαιωμάτων γυναικών και των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και στο δικό μας εδώ οίκο που δεν είναι πάντοτε σύμφωνοι και δεν ε, θέλουν να στηρίξουν. Δεν είναι το μόνο μας πρόβλημα ο Τραμπ. Την περασμένη εβδομάδα ψηφίσαμε έναν πρόεδρο εδώ, ο οποίος θα έλεγα ότι έχει κάποια προβλήματα στον τρόπο τον οποίο ε, τοποθετείται απέναντι στους ΛΟΑΔ. Επομένως δεν είναι μόνο θέμα της ε, πέρα όχθης του Ατλαντικού, είναι και δικό μας θέμα και δικό μας πρόβλημα Πώς λοιπόν μπορείτε εσείς να χρησιμοποιήσετε το καλό σας παράδειγμα ώστε τα θέματα πραγματικής ισότητας να υποστηριχθούν και να υλοποιούνται στην πραγματικότητα γιατί έχει σχέση με τις ευρωπαϊκές αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σας ευχαριστώ κύριος Μάρτιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ Υπουργέ για την τοποθέτησή σας. Σήμερα είναι η πρώτη μου συμμετοχή σε αυτήν εδώ την Επιτροπή Γυναικών και κατέφθασα ενθουσιασμένος γιατί περίμενα να δω μια αίθουσα γεμάτη άνδρες που θα μάχονται υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών. Γιατί τα δικαιώματα των γυναικών δεν είναι μόνο ιστορία, θέμα των γυναικών, είναι θέμα όλων μας. και ήθελα δύο σημεία, σε δύο σημεία να αναφερθώ, Υπουργέ. Γνωρίζω τη θέση της χώρας σας, αλλά έχω ακούσει και τη δική σας. Εισαγωγικά είπατε ότι πρέπει να προστατεύσουμε το κεκτημένο των ευρωαϊκών δικαιωμάτων. Και πρέπει να μην ξεχνούμε και το κεκτημένο σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και του δικαιώματος στην έκτρωση στην πρόορη διακοπή της κοιήσεως. Βλέπουμε τι συμβαίνει και στην Ήπειρό μας, βλέπουμε τι συμβαίνει στην Πολωνία, βλέπουμε τις διάφορες ε, εκδηλώσεις pro-life που διοργανώνονται και στη δική μας χώρα διάφορα συντηρητικά κέντρα υπόσχονται να ξαναθέσουν το θέμα της έκτρωσης. Τα θρησκευτικά θέματα έχουν επανέλθει και τοποθετούμαστε ε, επικρίνοντας εγκληματικά τις θέσεις ε, που είναι φιλικές προς την έκτρωση. Εγώ είμαι νεαρός πατέρας και βλέπω ότι υπάρχουν διάφορες αντιδραστικές πιέσεις που θέλουν να απαγορεύσουν από την μικρή μου κόρη να μπορέσει να αποφασίσει ελεύθερα επί του σώματός του στο μέλλον. Και είναι, θεωρώ, η κόρη μου ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του δράματος που θα μπορούσε να είναι μια πραγματικότητα δυστυχώς για πολλές γυναίκες. Επομένως όταν πισωγυρίζουμε σε σχέση με δεσμεύσεις και υποσχέσεις που έχουμε ακούσει, τι πρέπει να κάνουμε. Σε παγκόσμιο επίπεδο ε, το 77% των ηγετών τοποθετούνται κατά των εκτρέωσεων και πολύ μεγάλο ποσοστό εξ αυτών είναι άνδρες βεβαίως. Δεύτερον, αυτή η συμφιλίωση της επαγγελματικής ζωής και της προσωπικής ζωής. Το αναφέρατε και σας ευχαριστώ. Η πραγματικότητα που ζούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι αν ήμουν πατέρας στην χώρα σας θα είχα δικαίωμα σε δύο ημέρες άδεια και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μηδέν μέρες παρά το γεγονό ότι προσπαθούμε να δώσουμε μαθήματα σε, στους άλλους. Να τι κάνουμε στην πραγματικότητα. Επομένως, το να μιλούμε για τα δικαιώματα, την ισότητα των ανδρών και των γυναικών, είναι το να μιλούμε και για τα δικαιώματα των ανδρών στα θέματα, για παράδειγμα, των, της γονικής άδειας. Σας ευχαριστώ και τον προτείνω για τις απαντήσεις σας, Υπουργέ. Ευχαριστώ. Δεν θέλει κάποιος άλλο το λόγο. Οπότε, κυρία Υπουργέ, παρακαλώ, απαντήστε στα ερωτήματα. Ναι, για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για το θέμα αυτό. Έχουμε αλλάξει και θέση ως κυβέρνηση από αυτού. Με την αλλαγή της κυβέρνησης βέβαια. Ε, σε ό,τι αφορά τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Είναι ένα σημαντικό μήνυμα βεβαίως. Εμείς θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για την ε, επικύρωση. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα την ορατότητα του θέματος των γυναικών στα Δυτικά Συμβούλια, εμείς ε, θα το πάμε αυτό στην CSW, αλλά και ως Προεδρία στο Συμβούλιο. Είναι αλήθεια αυτό που ελέγχθη από την κυρία Ward για την πραγματική ισότητα μεταξύ των δύο φύλων που πρέπει να είναι πιο συμπεριληπτική ε, δεν μπορεί να αφορά μόνο τα δικαιώματα των γυναικών αλλά και την πραγματική ισότητα μεταξύ των φύλων. Θα έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να το ζητήσουμε αυτό στη διάσκεψη που θα οργανωθεί τον ερχόμενο μήνα. Τώρα τέθηκαν κάποια ερωτήματα νωρίτερα για τους στόχους ε, ε, σχετικά με το gender mainstreaming. Εμείς θέλουμε να προωθήσουμε την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Θέλουμε να εφαρμοστεί το mainstreaming σε αισθήματα φύλου ε, στην στρατηγική 2020 την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, ε, την ισότητα και το που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την επικύρωση της σύμβασης ε, της Κωνσταντινούπολης. Αυτή είναι η στόχη της ομάδας ψηλού επίπεδου που θα συνέλθει 1 και 2 Φεβρουαρίου. Και βέβαια υπάρχει και διάσκεψη για τη βία, τη διαμφιλική. Ε, θα συζητήσουμε τα αποτελέσματα από το Ινστιτούτο από το θεμελιώδες, ε, θεμελιώδη υπηρεσία, την υπηρεσία για θεμελιώδη δικαιώματα, συγγνώμη, ε, θα ανταλλάξουμε στοιχεία για βέλτιστες πρακτικές και θα δούμε ε, ποιες είναι οι πρακτικές στα διάφορα κράτη-μέλη, σε ό,τι την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και τις υπηρεσίες. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι η παρουσία των ανδρών εδώ δεν είναι τόσο εμφανής. Ε, συχνά, συχνά σε διασκέψεις μιλάνε και τις γυναίκες, ε, ε, μιλάω και λέω, εδώ μη, όμως προσπαθώ να, να πείσω άτομα που είναι ήδη πεισμένα. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερους άντρες όπως είπατε και τα αισθήματα που θέσατε βεβαίως θα πρέπει να απασχολούν τους άντρες όσο και τις γυναίκες. Οι, γυναίκες, άντρες έχουν συζύγους, έχουν κόρες, αδερφές, μητέρες. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε λοιπόν ως κοινωνίες, θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι οικογένειες και το πρίσμα της γυναίκας και το πρίσμα του άντρα. δεν μπορούμε να πούμε ότι, ξέρετε, οι γυναίκες να πούνε έχουμε τα προβλήματα και έχουμε και αυτές τις λύσεις. Ε, πρέπει να πούν και οι άντρες ποιες λύσεις βλέπουν. Είναι σημαντικό να έχουμε λοιπόν και τις δύο προοπτικές όταν προετοιμάζουμε πολιτικές για τη βελτίωση της διαβίωσής μας. Είστε, είστε βουλευτές, όπως και εγώ, και καθημερινά ε, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα τα, τα καθημερινά των ανθρώπων. Και πρέπει να μπορέσουμε αυτά να τα μετατρέψουμε σε νομοθεσίες. Και αν δεν μιλήσουν οι ίδιοι άντρες, οι ίδιες γυναίκες ε, ε, για αυτά που συζητούν μεταξύ τους ε, ε, στο τραπέζι είτε μιλάνε για την υγεία τους είτε μιλάνε για την ανεργία ε, για τα που τους απασχολούν ε, δεν πρόκειται να δημιουργηθεί αυτή η διασύνδεση που χρειάζεται μας χρειάζεται τόσο μεταξύ των πολιτών και των θεσμών το είδαμε πέρυσι με το Brexit υπάρχει ένα χάσμα ε, δεν βλέπουν ποια είναι η σημασία αυτών που συζητάμε εδώ. Νιώθουν ότι δεν έχουν θέση εδώ. Ε, δεν καταλαβαίνουν τι συζητάμε. Ε, ως βουλευτές εμείς και εσείς ως ευρωβουλευτές ε, πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε έτσι ώστε η καθημερινότητα των ανθρώπων ε, να ληφθεί υπόψη διότι αυτό είναι η κοινωνική βάση για την Ευρώπη. Εάν δεν αστροδιαβαθούν οι άντρε αυτά που λένε οι γυναίκε και τούμπαλιν, ε, και αν δεν αναζητήσουμε λύσεις από κοινού, λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ε, στις γειτονιές μας, ε, στις κοινωνίες μας, Λέμε συχνά πως ε, σε κάποια κράτη-μέλη όπως το δικό μου ε, πρέπει να αυξηθεί η γονιμότητα. Από την άλλη λέμε ότι σας θέλουμε στην αγορά εργασίας, ε, ε, επενδύουμε στην εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά χάνονται οι επενδύσεις αυτές γιατί δεν υπάρχουν δομές για τις οικογένειες για να μπορούν να κάνουν και τα δύο και να έχουν παιδιά και να μπορούν να ε, εργαστούν ικανοποιητικά και να το κάνουν αυτό ε, με την ηρεμία, με την γαλήνη μια ασφάλειας, ε, ότι μπορούν να τα κάνουν και τα δύο. Η κοινωνία προχωράει εφόσον δημιουργήσουμε εμείς τις απαραίτητες δομές για τις οικογένειες και να μπορούν να το κάνουν αυτό. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους και στην οικογένειά τους αλλά και στον χώρο εργασία τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερος που ήρθατε σε αυτή τη συνάντηση και που παρουσιάσατε τις προτεραιότητες της Μαλτέζικης Προεδρίας. Θα ήθελα πραγματικά ε, να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία για την Προεδρία σας. Ελπίζουμε να φέρει αποτελέσματα θα τα ξαναπούμε σίγουρα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Για άλλη μια φορά σας εύχομαι κάθε επιτυχία. svarstėm visus mūsų klausimus, noriu pasakyti. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τα σημεία της ημέρας διάταξης για σήμερα. Η επόμενη συνάντηση θα λάβει χώρα στις 6 Φεβρουαρίου, στις 3 το απόγευμα. Σα ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Και τώρα μια σύντομη συνάντηση των συντονιστών. Ευχαριστώ.